Bien, chers collègues, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, veuillez. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ να λάβετε τις θέσεις. Euh, assez rapidement, puisque le commissaire Barnier euh, est disponible pour euh, une heure avec nous. Ας αρχίσουμε, διότι έχουμε ήδη μαζί μας τον Επίτροπο κύριε Μπανέ. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ για αυτή την ακρόαση που κάνουμε τις εργασίες της Επιτροπής μας μετά από το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, στο οποίο συζητήθηκαν θέματα ασφαλείας και άμυνας, κοινή πολιτικής ασφαλείας και άμυνας, η task force που σύστησε η Επιτροπή με τον συνάδελφό σας, τον κύριο Ταγιάννη, με τον οποίο θα έχουμε μια ακρόαση αργότερα, πρέπει να επεξεργαστεί διάφορα θέματα τα οποία αφορούν την Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία και θα ακούσουμε με προσοχή αυτά τα οποία έχετε να μας πείτε για τις εργασίες αυτής της Task Force, αυτής της ομάδας εργασίας. Βεβαίως, μας απασχολεί η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών αμυντικών βιομηχανιών, αλλά θέλουμε οπωσδήποτε η ανταγωνιστικότητα αυτή να γίνει στα πλαίσια ενός στρατηγικού σχεδίου για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για βιομηχανία η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική για την Ευρώπη, αλλά είναι μεγαλύτερες οι φιλοδοξίες μας. Δηλαδή αυτό το οποίο επαναλαμβάνονται στις διάφορες εκθέσεις που εγκρίνονται με μεγάλη πλειοψηφία παρά το γεγονό ότι κάποιοι δεν σημαίνει την απόψή μα να δώσει στρατηγική αυτονομία για να εξαρτησία θέματα άμυνα στην Ευρώπη. Και βεβαίως είμαστε σε συχνή επαφή με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Θα μας πείτε κι εσείς πώς διαμορφώνεται στα πλαίσια της Tax Force αυτής η συνεργασία των, ε, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Μέχρι τώρα ξέρουμε ότι δεν τα είχε ίσως και πάρα πολύ καλά η Επιτροπή με τα θέματα άμυνας και χαιρετίζουμε το ότι είστε εδώ στην υποεπιτροπή μας και ελπίζουμε ότι μετά από την ανταλλαγή απόψεων που θα έχουμε θα μπορέσουμε να έχουμε πιο σαφή άποψη για αυτά τα οποία διαμήφθησαν κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου, στην οποία δεν ζητήθηκε η παρουσία μα, αλλά φαντάζομαι ότι και επί αυτού του θέματο θα υποβάλουν κάποιε προτάσει οι συνάδελφοι, διότι πρόκειται για θέματα σημαντικά. Σημαντικά είναι τα θέματα τα οποία ασχολείται. Το θέμα της πολιτική στο Μαλί και όλα αυτά είναι θέματα και εξωτερική πολιτική και άμυνας θέματα εξαιρετικά σημαντικά και για τα κράτη μας και για τους πολίτες της Ευρώπης. Σας δίνω το λόγο αμέσω, κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την υποδοχή σας και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους παρευρισκόμενους για την προσοχή. Δεν είναι η πρώτη φορά που παρίσταμε στις εργασίες της Επιτροπή, σα, τη Επιτροπή που ασχολείται με θέματα άμυνα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τον προκάτοχό σα. Είχαμε συναντηθεί το 2006, είχα παρουσιάσει τα συμπεράσματα της εργασίας που είχα κάνει εκτός Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική προστασία. Ε, μου το είχε αναθέσει την εργασία αυτή ο πρόεδρος Μπαρόζο για να μπορέσουμε να συστήσουμε την ευρωπαϊκή δύναμη της πολιτικής προστασίας. Και όσοι με γνωρίζουν ξέρουν ότι τα θέματα αυτά με ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Όχι διότι εγώ έχω υπάρξει εδώ και χρόνια υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας, αλλά ότι είχα την τιμή να προεδρεύσω στα πλαίσια της ε, Ευρωπαϊκής Σύμβασης, της ομάδας εργασίας που ασχολήθηκε με θέματα ευρωπαϊκής άμυνας. Και από αυτή την ομάδα, εάν θέλετε, προέκυψε το κεφάλαιο που αφορά στη συνθήκη της Λισαβόνας όλα τα θέματα τα οποία αφορούν την άμυνα. Πρόκειται λοιπόν για τα πορίσματα της ομάδας εργασίας της οποίας προείδευε. Εδώ μιλούμε για την πρόσφατη πολιτική στον ευρωπαϊκό τομέα για τις πρώτες γενικές γραμμές της ΚΕΠΑ. Ας αρχίσουμε από το 1991 που είχαμε τις πρώτες ε, ε, στρατιωτικές και μη στρατιωτικού χαρακτήρα επιχειρήσεις που είχαν αρχίσει κάποια χρόνια πριν. Μιλούμε για μια πολιτική η οποία δεν είναι κοινοτική και δικαίω είπε ο Πρόεδρος ότι η παρουσία ενός Ευρωπαίου Επιτρόπου στην Επιτροπή σας είναι κάτι το καινούριο. Κάτι το πρόσμενο θα έλεγαν. Γιατί όμως. Μπορεί να γίνει κατανοητή και να είχαμε και χρήσιμη η παρουσία του Επιτρόπου που ασχολείται με αυτά τα θέματα. Διότι εμείς έχουμε μια άλλη εντελώς οπτική γωνία για αυτή την πολιτική σε σχέση με τις άλλες κοινωτικέ πολιτικές. Πρόκειται για μια νέα πολιτική στην ε, οποία μπορούμε να πάμε πάρα πολύ μακριά θα πρέπει να είμαστε για αυτή την πολιτική άμενας αμερόληπτοι, αντικειμενικοί, διότι πολλές φορές παρά το γεγονός ότι είναι κάτι το πρόσφατο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να πω ότι επικρίνεται. Πρέπει να πω ότι έχουμε 27 διαφορετικά συστήματα στρατιωτικά, ειδικά. Έχουμε μεταξύ των κρατών μελών ε, διάφορα ουδέτερα στρατιωτικά κράτη, αν θέλετε οι αμυντικέ βιομηχανίες είναι διαφορετικές, οι παραδόσεις είναι διαφορετικέ και έχουμε να κάνουμε μια πολιτική κατεξοχήν ε, διαφορετική για κάθε χώρα. Είμαι παρόλα αυτά πεπισμένος ως πολιτικός και ως επίτροπος ότι είναι η κατάλληλη στιγμή, είναι επίγουσα σημασία να δώσουμε μια νέα όθηση στην ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας και ασφάλεια. Πρώτα απ' όλα διότι όπως βλέπετε υπάρχουν νέες απειλές δεν βρίσκονται γεωγραφικά πολύ μακριά από την δική μας την Ήπειρο και αναφέρομαι ιδιαίτερα στην Αφρική και πρόκειται για απειλές που μας αφορούν άμεσα μας τους Ευρωπαίους. Ο δεύτερος λόγος είναι διότι σε επίπεδο κοινοτικού προϋπολογισμού τον οποίο ασχολείστε εσείς, καθώς και με κάθε εθνικό προϋπολογισμό στη χώρα σας, βλέπετε ότι υπάρχουν προβλήματα και περιορισμοί οικονομικοί που, εάν Θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι και να έχουμε δυνατότητες θα πρέπει να χειριστούμε θέτοντας από κοινού τους πόρους που διαθέτουμε στον τομέα αυτό, καθώς και τον τομέα της έρευνας, Φερρυπίν. Επίσης, στην ετήσια έκθεση έγινε λόγος για τις νέες στρατηγικής σημασίας προτεραιότητες των Ηνωμένων Πολιτειών των συμμάχων μας, για τους οποίους θεωρούμε πολλούς σημαντικούς, παρά το γεγονός ότι θέλουμε να είναι ισοσκελισμένη αυτού του είδους η ισορροπία μεταξύ ΕΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ε, έχουμε επιτύχει αυτό το αποτέλεσμα προς το παρόν και άκουσα τον αντιπρόεδρο, τον ΙΠΑ, τον Τζο Μπάιντον στο Μόναχο, μας είπε σε εμάς τους Ευρωπαίους ότι η Ευρώπη σε θέματα ασφαλεία για τους Αμερικανούς είναι ακρογωνίως λίθος. αλλά πρέπει να επορμιστείτε τις ευθύνε σας ως Ευρώπη. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτό το νέο ε, γεωπολιτικό πλαίσιο με στο οποίο θα πρέπει να κινηθούμε και να δώσουμε νέα όθηση σε αυτή την ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας και να επομιστούμε τις ευθύνες μας για την δική μας ασφάλεια. Ε, υπάρχουν διάφορα μέσα Ανέφερα τη συνθήκη της Λισαβόνας, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας και εάν υπάρχει πολιτική βούληση, πράγμα το οποίο επιθυμώ, θέλω να πραγματοποιηθεί, αλλά πολλές φορές βλέπω να υπάρχουν σε επίπεδο κρατών μελών ενδιασμοί και αδυναμίες. Αν υπάρχει λοιπόν η πολιτική βούληση, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Και από αυτού του σημείου, δεδομένου ότι πρόκειται για την ε, προπαρασκευή μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύω ότι μπορεί να προσδώσει μία προστιθέμενη αξία στο θέμα αυτό. Έχει κάτι το χρήσιμο να προσφέρει. Αν δούμε τα πορίσματα του Συμβουλίου Άμυνας του Δεκεμβρίου 2012 και αν θέλουμε να προετοιμάσουμε με αποτελεσματικό τρόπο το αντίστοιχο ε, Συμβούλιο φέτος το Δεκέμβριο, και εδώ και πολύ καιρό, όπω υπενθύμισε ο πρόεδρο Ντοζό, υπό την όθηση του πρόεδρου Βον Ρομπάη, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ελπίζω ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο χωρί να υπάρξει ε, η οικονομική κρίση μεγάλη, η οποία θα μας αποπροσανατολίσει, κυρίως θα προσδώσει την πρώτη προτεραιότητα στην ευρωπαϊκή πολιτική άμυνα. Θέλουμε λοιπόν να προετοιμαστούμε κατάλληλα έω τότε. Και σε τρεις κυρίως για τρία μεγάλα θέματα. Πρώτα απ' όλα, να μπορέσουμε, αν είναι δυνατόν, να θέσουμε από κοινού τα μέσα τα οποία διαθέτουμε στον στρατιωτικό και πολιτικό τομέα για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις και τις απειλές. Πρόκειται για εργασία που γίνεται από την διπλωματική ε, υπηρεσία της Ευρώπης, από την συνάδελφό μου την κυρία Άστον. Αλλά υπάρχει σχέση με το θέμα των δυνατοτήτων που διαθέτουμε. Και εδώ έχει δεσμεύσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, το πρώτο αυτό σκέλος που ανέφερα είναι ε, θέμα αρμουδιότητος διακυβερνητικών των κυβερνήσεων και των εκπροσώπων των κυβερνήσεων. Δεύτερο σκέλος. Συνεργασία, pooling and sharing. Θέτω το μέσο από κοινού και μοιράζομαι για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις ε, δυνατότητες των κρατών μελών και από την άποψή μου, κατά την άποψή μου, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να κάνουν μεταξύ τους οι Ευρωπαίοι. Το πρώτο λοιπόν ε, βήμα λοιπόν για να μπορέσουμε να θέσουμε από κοινού τα μέσα που διαθέτουμε και να ενεργήσουμε είναι να δούμε τι θα κάνουμε με τις ε, αγορές στον τομέα των, ε, της ε, αμυντικής βιομηχανίας. Πρέπει να γίνει πιο ανταγωνιστική και να μπορούν να παρέχουν στους Ευρωπαίους τους εξοπλισμούς, τα μέσα που χρειάζονται για την δική τους ε, ασφάλεια και άμυνα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εδώ λοιπόν μπορεί να είναι χρήσιμη, δεδομένου ότι έχει τις ε, κανονιστικές δραστηριότητες και διαθέτει την ε, πραγματογνωμοσύνη που χρειάζεται για κανόνες για προδιαγραφές και έχει και τα κατάλληλα οικονομικά προγράμματα στα πλαίσια των διαρθρωτικών ταμείων μεταξύ άλλων. Γι' αυτό κυρίες και κύριοι με τον συνάδελφό μου, τον κύριο Ταγιάννη, μας απασχολούν και ασχολούμεθα με τα θέματα αυτά, όχι μόνο στα πλαίσια αυτών των δύο μέσων του πακέτου άμυνας που έχουμε, τις δύο οδηγίε δηλαδή, για να εφαρμοστεί αυτή η πολιτική, διότι πέραν από την ε, μεταφορά και αυτών των οδηγιών σε κάθε εθνικό δίκαιο και στην θέση της σε ισχύ, για να προετοιμαστούμε σωστά και να ενεργήσουμε σωστά, γνωρίζουμε ότι χρειάστηκε πολιτική βούληση. Και ο Αντώνιο Ταγιάννη, που θα έρθει στην Επιτροπή σας, την οποία θα έχετε μια κρόση σε μια επόμενη συνεδρίασή σας, δημιουργήσαμε μία task force στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη συνδρομή περίπου 10 γενικών ε, διευθύνσεων που θα σας απαριθμίσω επιγραμματικά. Πρώτα απ' όλα, εσωτερική αγορά των ε, αμυντικών βιομηχανιών. Μελετούμε τις δράσεις για να έχουμε μεγαλύτερο άνοιγμα την αγορά και να βελτιώσουμε την κατάσταση της βιομηχανίας αυτή δίδοντας την σωστή ερμηνεία στο άρθρο 346 των συνθήκων που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό το οποίο θέλουμε κυρίως είναι οι διάφορες γενικές διευθύνσεις να δώσουν συντονισμένη συνεκτική ερμηνεία του άρθρου αυτού 346. Δεύτερο θέμα, η βιομηχανική πολιτική άμυνας πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτές τις χιλιάδες επιχειρήσεις, κυρίως τις ΜΜΕ που εργάζονται στον τομέα της άμυνας, πώς μπορούμε να τις βοηθήσουμε να κάνουν αναδιαρθρωσίες, πώς να αρχίσουν νέες επιχειρήσεις, νέες startup, πώς να διευκολύνουμε διάλογο σε όλους τους ε, τομείς που συμμετέχουν για την ε, ανταγωνιστικότητα του τομέα αυτού, κοινά στάνταρ, κοινοί κανόνες, και αυτά είναι θέματα αρμοδιότητάς μου για την ε, ασχολούμαι θέματα της ιστορικής αγοράς και για το απόλυτο στον τομέα αυτό. Τρίτος τομέας, η ενέργεια. Γνωρίζουμε ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι ο τομέας του δημοσίου που χρησιμοποιεί τις μεγαλύτερες ποσότητες ενέργειας. Και θέλουμε να είμαστε αποδοτικοί και οικονομικοί σε θέματα ενέργειας. Άρα, προς συμφέρον τους, για οικονομικούς λόγους και οικολογικούς θα είναι να μειώσουν την ενέργεια που καταναλώνουν. Πιστεύουμε ότι στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Ενέργεια έχει εδώ την κατάλληλη θέση της και η ενεργειακή πολιτική στον τομέα της έρευνας. Τέταρτο θέμα, δυνατότητες διτές. Στο παρόν πλαίσιο της ε, ασφάλειας, οι δυνάμεις ασφαλείας χρειάζονται ε, παρεμφερείς δυνατότητες και παρεμφερή μέσα, κυρίως όταν συμμετέχουν στην ίδια αποστολή ή επιτόπου έχουν άμεση συνεργασία όπως, ε, για να φέρω παράδειγμα, την προστασία των ε, εξωτερικών συνόρων, την εποπτεία των θαλασσίων συνόρων, τη διαχείριση κρίσεων ή την ε, σύνδρομη και αρρωγή σε περίπτωση καταστροφής. Όπως ξέρετε, κάναμε μια εργασία για την ενίσχυση πολιτικής προστασίας και την θέση από των μέσων που διαθέτουμε. Κάνουμε λοιπόν πολιτικές ασφάλειας για θέματα μη στρατιωτικών οστολών και Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης προσπαθεί να δει όλα τα θέματα που αφορούν τις ε, δυνατότητες που έχουμε. Προς το παρόν, με τι ασχολούμεθα, με τις ε, δυνατότητες των κρατών μελών αλλά αν πρέπει να σας μιλήσω με ειλικρίνεια, είμαι μεταξύ αυτών που πιστεύουν ότι αναμφίβολα και θα πω τη γνώμη μου ανοιχτά, πρέπει να είμαστε πιο ευφυείς, πιο αποτελεσματικοί και στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε κάποιες δυνατότητες να τις εκμεταλλευτούμε εμείς οι ίδιοι για να ανταποκριθούμε σε θέματα ασφαλείας. Με τον Καλλιλέο επιλέξαμε στην Ευρώπη για την ε, ε, πλοήγηση ε, το σύστημα αυτό και διερωτώμε με δεν θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως πρότυπο αυτό που κάναμε εδώ με τον Καλλιλέο και για άλλους στρατηγικούς τομείς. Όχι μόνο για το στρατιωτικό τομέα, αλλά για τον ασφάλεια ή για μη επανδρομένα αεροσκάφη, για την εποπτεία των συνόρων ή για πλοία νοσοκομεία ή για μεγάλα αεροσκάφη μεταφορικά, μεταγωγικά, ώστε να μπορεί να ενεργεί μόνη της η Ευρώπη και να μπορεί κάποια εξοπλισμό να τον αποστέλει σε κάποιες χώρες χωρίς να χρειάζεται βοήθεια του. Αυτά είναι θέματα συνολικής σφαιρικής ασφάλειας και το είπα στην έκθεσή μου για την πολιτική προστασία. Χώρες μας όπως η Ισπανία, η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία αντιμετωπίζουν πολλές φορές προβλήματα ρήπανσης των υδάτων των θαλασσών και θα πρέπει να διθέτουμε για σε περιορισμένο ε, μέγεθος βεβαίως να έχουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό για να μπορούμε να προστατεύουμε τις, χώρες, τις ακτές μας και τις Τελικά όλα αυτά είναι και θέματα οικονομικών πόρων και πολιτικών επιλογών και βούλησης βεβαίως. Το διάστημα, το επόμενο θέμα θέμα για το οποίο είναι υπεύθυνο ο συνάδελφος Ταγιάννη. Επίσης εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν ε, τομέα ο οποίος είναι διπλόζητος, αν θέλετε. Πρέπει να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε με ευφύ τρόπο όλες τις συνέργειες μεταξύ του ε, πολιτικού και του στρατιωτικού τομέα. Και δεδομένου ότι μιλούμε για το διάστημα, θα παραμείνω όχι στον ουρανό. Δεν θα πάω πολύ ψηλά υπάρχουν τομείς στους οποίους θα μπορούσε ε, στην υπηρεσία των κρατών μελών να χρησιμοποιήσει και τις κανονιστικές της ε, αρμοδιότητες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυρίως αναφέρομαι στην αεροπλοεία, κυρίως για τις στρατιωτικές πτήσεις, τις πτήσεις αμυντικού χαρακτήρα. Έκτο θέμα είναι το θέμα της έρευνας, όπως και για το διάστημα τα προγράμματα της έρευνας τα οποία χρηματοδοτούμε ασχολούνται με μη στρατιωτικές ε, έρευνες και χρήσεις. Αλλά περιλαμβάνουν όμως κάποιες διπλής φύσης ε, πλευρές. Και εκεί πρέπει να προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες συνεργασίας. Και τέλος έχουμε το θέμα του εμπορίου. Εκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλύπτει θα έλεγα και έχει ευθύνη για όλες τις εμπορικές συναλλαγές μη στρατιωτικής φύσης. Τα θέματα των αμυντικών <clears throat> προμηθειών δεν καλύπτονται από τις αρμοδιότητές μας, δεν τίθεται λοιπόν θέμα κοινή δράση. Το θέμα όμως το οποίο τίθεται είναι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο έτσι ώστε να βελτιωθεί το περιθώριο προόδου και δράσης και πρόσβασης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις αμερικανικές ας πούμε αγορές και σε τρίτες αγορές επίσης. Αυτή τη στιγμή αποφασίσαμε ε, να καταργήσουμε τα αντισταθμιστικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Αυτό είναι το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμεθα και προσπάθησα να σας περιγράψω τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει και μπορεί να είναι χρήσιμη σε μια μελλοντική κοινή ή ενιαία αγορά των αμυντικών βιομηχανιών. Μια τελευταία λέξη για τα θέματα ακριβώς των αμυντικών βιομηχανιών. Ανήκουν στην ευρωπαϊκή βιομηχανία βέβαια, η οποία σε αυτή τη φάση είναι θα έλεγε κανείς ιδιαίτερα έθραυστη και σε σχέση με άλλες χώρες μάλιστα ε, χάνει κάποια τμήματα της αγοράς. Ό,τι κάνουμε εμείς σαν Επιτροπή σε συνεργασία με εσά έχουν σαν στόχο την βελτίωση του οικοσυστήματος θα έλεγα μέσα στο οποίο δημιουργούν και εξάγουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Δύο βασικές πολιτικές τις οποίες ε, ε, στηρίζουμε με την δική σας φυσικά σύμφωνη γνώμη. Το είναι πολιτική μας το θέμα της εσωτερικής αγοράς. Ε, με δέκα άλλους επιτρόπους έχουμε συντάξει μια ατζέντα για την ανάκαμψη θα έλεγα της οικονομίας, τα Single Market Acts 1 και 2 περιλαμβάνονται 55 προτάσεις επιμέρους με στόχο την βελτίωση της εσωτερικής αγοράς, εξυπηρετώντας όλες τις βιομηχανικές δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων και την αμυντική βιομηχανία. Όταν μιλάμε για το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, όταν μιλάμε για το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Προϊόντων, Ξέρετε ότι χτες ε, υπήρξε μια πρώτη συμφωνία 25 χωρών ε, για το πρώτο ε, ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, το οποίο από του χρόνου θα κάνει 2.500 ευρώ και όχι 20.000 που κάνει σήμερα. Όταν μιλάμε σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ηλεκτρονική υπογραφή των συναλλαγών στο διαδίκτυο, καλύπτουμε τις ανάγκες όλων των ευρωπαϊκών βιομηχανιών, μεταξύ των οποίων και των αμυντικών βιομηχανιών. Έτσι λοιπόν, βλέποντας τι έχουμε να κάνουμε, βλέπουμε ότι εδώ και λίγο καιρό σε συνεργασία με τον κύριο Ταγιάννη προσπαθούμε να καταθέσουμε μία πρόταση για ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική, εφόσον το επιθυμούν τα κράτη-μέλη. Ο Ταγιάννη, σε συνεργασία με κάποιους εμπειρογνώμονες, οδηγήθηκε στον κατάλογο 7-8 τεχνολογιών κλειδιά, στα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύει να χάσει την αυτονομία της και αυτά όλα έχουν πολύ μεγάλη σημασία, όχι μόνο για την αμυντική βιομηχανία, αλλά για την ασφάλεια της Ευρώπης. Λοιπόν, δεν θα πρέπει να κρατήσουμε μία κάποια αυτονομία στην Ευρώπη, αντί να την αγοράζουμε κάθε φορά από τους Αμερικανούς, τους Ιάπωνες ή τους Κινέζους. Αυτά πρέπει να κάνουμε. Δεν ξέρω αν θα το καταφέρουμε αυτό αλλά κάνουμε προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτών των κομβικών τεχνολογιών. Στα πλαίσια της ενίας αγοράς λοιπόν, κάτι το οποίο ενδιαφέρει και τις αμυντικές βιομηχανίες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ λέει και ο κύριος Ντανζό πριν δώσω το λόγο στους συναδέλφους να πω ότι στην παρέμβασή σας άκουσα κάποιες λέξεις κλειδιά. Κάποιες λέξεις που δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατανοεί ότι στα θέματα της βιομηχανίας της άμυνας δεν μιλάμε για βιομηχανικούς τομείς οι οποίοι είναι ίδιοι με όλους τους άλλους. Οι τεχνολογίες διαφέρουν και ο στρατηγικός χαρακτήρας των ε, πολιτικών διαφέρει. Ως εκ τούτου λοιπόν η αγορά αυτή αποκτά μια νέα διάσταση, μια διάσταση την οποία θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη εφόσον θέλουμε να προχωρήσουμε στις απαιτούμενες ρυθμίσεις. Ο κύριος Γκάλα, συντονιστής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Ήθελα να περιμένω λίγο να φορέσετε τα ακουστικά σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ θερμά για την παρουσίασή σας. Οι συναντήσεις αυτές ε, παρακολουθούνται με ανοιχτό πνεύμα από το ΕΛΚ και συμφωνούμε ότι θέλουμε ανταγωνιστική βιομηχανική βάση στην Ευρώπη, τεχνολογική βάση και μεταξύ άλλων να κρατήσουμε ζωντανές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας. Αν ξεπεραστούν οι εθνικοί εγωισμοί σε αυτό το τομέα, θα ακολουθούμε σωστό δρόμο. Ε, στην ειδική ομάδα για την ε, άμυνα που συστήσατε με τον συνάδελφό σας κύριο Ταγιάννη, κάνατε μια καλή επιλογή. Ήταν καλό το ότι συστάθηκε αυτή η ειδική ομάδα. Ε, σε ό,τι αφορά το πακέτο άμυνας έπρεπε η οδηγία για τις ε, αμυντικές προμήθειες και τα προϊόντα άμυνας θα έπρεπε οι δύο οδηγίες να εφαρμοστούν. Αυτό έγινε. Σε ποιο βαθμό ακολούθησαν τα κράτη-μέλη το δρόμο της εφαρμογής των δύο οδηγιών. Αυτό θα με ενδιαφέρε να μου το πείτε. Και επειδή είστε ε, αρμόδιος για την αγορά, βλέποντας τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας, παρακολουθώ ότι έχει ένα μεγάλο τμήμα που αναφέρεται στην αγορά. Κανονικά θα έπρεπε αυτό το κομμάτι από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας για την αγορά θα έπρεπε να πάει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί ε, υπάρχει σε δύο διαφορετικούς ε, τομείς και επίπεδα. Επίσης, ε, στην περασμένη ετήσια έκθεση του κ. Μπρόκ ζητούμε από το, του χρόνου στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο ο οργανισμός άμυνας να χρηματοδοτείται από, την, από τον ενωσιακό προϋπολογισμό και καλούμε την Λέδη Άστο να υποβάλει σχετικές προτάσεις. Γνωρίζετε κάτι εάν προτίθεται η κυρία Άστο να υποβάλει σχετική πρόταση ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, ούτως ώστε το... τα... οι λειτουργικές δαπάνες ε, να... του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας να χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, αλλιώς θα παρέμενε υπόθεση των κρατών μελών. Ε, νομίζω ότι χρειάζεται αυτή η κοινή προσέγγιση. Εδώ στο Κοινοβούλιο εδώ και καιρό ζητούσαμε με βάση τις εξελίξεις να υπάρξει λευκή βίβλος για την ασφάλεια και την άμυνα με βάση ε, μιας defense review, μιας ανασκόπησης της άμυνας και να δούμε ποια είναι τα προϊόντα στον τομέα των εξοπλισμών που θα πρέπει να προωθηθούν, τι πρέπει να γίνει ούτως ώστε να λάβουμε υπόψη μας τα νέα δεδομένα στον τομέα της ασφάλειας και πώς θα μπορούσαμε να ορίσουμε τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Βλέπετε τη δυνατότητα αν υπάρξει τέτοια λευκή βίβλος η Κομισιόν να έχει να κάνει μια σημαντική συμβολή. Αυτά είναι σοβαρά θέματα για μένα. Από την άλλη καλό θα ήταν να μπορούσαμε να προχωρήσουμε στην consolidation of demand ή την εναρμόνιση της ζήτησης ή την ε, δρέωση ε, και εξυγίαση της ε, ζήτησης. Αν έχουμε 10 μοντέλα διαφορετικά του Tiger, θα βλέπαμε αλλιώ το θέμα της συμπατότητας ή της τιμής. Καλό θα ήταν λοιπόν και η Κομισιόν να ασκήσει επιρροή στα κράτη-μέλη τους, ώστε κάποιες πρακτικές να αλλάξουν. Και θα πρέπει να έχουμε και προσανατολισμό προς την βιομηχανία. Αλλιώς ε, θα έπρεπε να ζητήσουμε από την βιομηχανία να έχει μόνο δύο μοντέλα και να το δεχτούν τα κράτη-μέλη αναγκαστικά. Πώς λοιπόν βλέπετε τη στάση των ε, κρατών μελών ε, θα δεχθούν τις προτάσεις σας και τις προσεγγίσεις σας που νομίζω ότι είναι σωστές και θα δράσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Έχουμε 20 λεπτά στη διάθεσή μας, γι' αυτό παρακαλώ στις ερωτήσεις σας να είστε σύντομοι για να μπορέσουμε να ακουστούμε όλοι. Ο κύριος Σοφοκλέους. Έχω παρακολουθήσει με προσοχή τα όσα έχετε πει και θα συμφωνήσω μαζί σας με τον τρόπο που έχετε παρουσιάσει, θα έλεγα, μια πρόταση ενημέρωση που κινήθηκε προς τρεις άξονες. Η πρώτη είναι η διαπίστωση ότι Υπάρχουν νέες απειλές ειδικότερα στην Αφρική και πρέπει να δοθεί μια νέα όθηση. Ο δεύτερος άξονας είναι οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν θα τις σχολιάσω παρά μόνο να υπογραμμίσω ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε έριξαν το βάρος προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για να λάβουμε τις ευθύνε μας. Και ο τρίτος άξονας είναι ο προϋπολογισμός. Η ερώτηση μου είναι εξή αναφορικά με τον προϋπολογισμό και τους κοινού πόρους που πρέπει να διατεθούν για την άμυνα ουσιαστικά. Υπάρχουν κάποια, κάποιο σχέδιο, υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πρόταση, γιατί όπως ξέρετε ο καυγάς όλος που γίνεται είναι για τα χρήματα, είναι πώς θα διατεθούν χρήματα. Ήδη είδαμε τι έγινε με τη μείωση του προπολογισμού και νομίζω ότι στο διατάφτα είναι να απαντήσουμε και να απαντήσει, αν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πολιτική πρόταση, ένα σχέδιο που θα επηρεάσει θετικά τις χώρες που συμμετέχουν να διαθέσουν βεβαίως τα μέσα αλλά κυρίως τα χρήματα. Υπάρχει κάποιος τρόπος. Merci, Madame Nates. Κύριε Νάιτς, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα είμαι σύντομη. Οι ερωτήσεις που θα ήθελα να θέσω είναι, θα έλεγα, μία προέκτηση αυτών που ήδη είπε ο κύριος Γκάλα. Θεωρώ ότι όλος παραδόξος οι δημοσιονομικές δυσκολίες οι οποίες σοβούν στις περισσότερες χώρες και στις οποίες ήδη αναφερθήκατε ανοίγουν ένα παράθυρο ευκαιρίες, ε, κάτι το οποίο σπάνια είχαμε συναντήσει στο παρελθόν. Κάτω από αυτές τις δημοσιονομικές πιέσεις, τα κράτη-μέλη δεν έχουν την δυνατότητα να προχωρήσουν εύκολα σε δαπάνες στον τομέα των στρατιωτικών ή των αμυντικό γενικότερα. Επανέρχομαι λοιπόν στο ερώτημα του κυρίου Γκάλερ. Εδώ δεν λειτουργούμε και κλεισμένων των θύρων και πρέπει να θέσω την ερώτησή μου. Θα μπορούσατε να μας πείτε αν έχουν υπάρξει κάποιες εξελίξεις στις αντιλήψεις και στις νοοτροπίες των κυβερνήσεων των κρατών μελών γύρω από τα θέματα αυτά. Κάτι το οποίο να ξεπερνάει δηλαδή την απλή οργάνωση κάποιων συναντήσεων ενδιαφέρουσων βέβαια όπως αυτή του Σαμαλό. Αλλά παρόλα αυτά κάτι το πιο συγκεκριμένο, κάτι το πιο απτό ε, πώς προχωρούν λοιπόν οι επαφές ανάμεσα στα κράτη-μέλη των κρατών μελών σε επίπεδο υπουργών και σε επίπεδο υπουργών στρατιωτικών. Ο κύριος Μπούτι Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στο non-paper της Κομισιόν διάβασα αυτά τα κενά ικανοτήτων είναι άμεση συνέπεια των δημοσιονομικών περιορισμών αυτό δεν με πείθει. Τα κενά στις ικανότητες που έχουμε σήμερα αποτελούν α, συνέπειες αποφάσεων που ελήφθησαν πριν από 10-20 χρόνια. Δηλαδή, οι σημερινοί δημοσιονομικοί περιορισμοί δεν έχουν σχέση με τα κενά. Πιστεύω όμως ότι οι δημοσιονομικοί περιορισμοί πρέπει παρόλα αυτά να ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη υπό την έννοια της ερώτησης κυρίας Νάιτς, δηλαδή ποια στρατηγική θα ακολουθήσουμε ε, σε σχέση με τη συνεργασία στο τομέα των ικανοτήτων. Αν δεν εδώ χρειάζεται απόφαση φιλόδοξη για μεγαλύτερο pooling και sharing, συνένωση και κοινή χρήση. Αλλιώς η αμυντική βιομηχανία στην Ευρώπη θα ε, οικοδομηθεί σε ολιστηρό έδαφος. Τώρα, για τις εξαγωγές εξοπλισμών πρέπει να προσέξουμε να μην είμαστε μονόπλευροι και να μην δούμε το θέμα μερκαντιλιστικά. Θα πρέπει να θέσουμε σοβαρά το ερώτημα πόσο έξυπνο είναι για την παγκόσμια σταθερότητα και ασφάλεια να ε, στείλουμε ευρωπαϊκούς εξοπλισμούς στην Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική με κίνδυνο ανάφλεξης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επίτροπε Μπαρνιέ, πάντα είναι μεγάλη χαρά να ακούμε τις απόψεις σας. Βεβαίως στην ε, ε, κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας ε, έχετε μεγάλη εμπειρία και οι προτάσεις σας είναι πολύ λογικές, ακούγονται εύλογες. Βεβαίως η πολιτική αυτή θα πρέπει να αναβαθμίσει την Ευρώπη ως παγκόσμιο παίκτη και δεν έχει τόσο σχέση με τις ανάγκες της άμυνας. Ερώτηση. Δέχεστε ότι η Κομισιόν φιλοδοξεί σταδιακά να κοινοτικοποιήσει την άμυνα. Δηλαδή είναι αυτή η κατεύθυνση που θέλετε να ακολουθηθεί και βλέπετε ότι κινούνται κάποια πράγματα εκεί. Λέτε ότι αντιμετωπίζουμε νέες απειλές. Είναι διαφορετικές από τις απειλές που αντιμετωπίζει το ΝΑΤΟ. Ακόμα και αν δούμε τις επεμβάσεις, τις ε, ε, πρώην ε, γαλλικές ε, περιοχές ενδιαφέροντος στην Κεντρική Αφρική βλέπουμε μεγάλη εμπλοκή των ΙΠΑ. Βλέπουμε ενισχυμένε προσπάθειες σε γειτονικέ χώρες, στο Μάλι, στον Νίγηρα και άλλες χώρες παρόμοιες. Και για να ανταποκριθούμε στις πολύ σοβαρές αυτές απειλές χρειάζεται προσπάθεια συμμαχική. Δηλαδή χρειαζόμαστε τις ΙΠΑ και άλλους ε, πρόθυμους ε, συμμάχους. Και είδαμε στην επέμβαση στη Λιβύη ότι κάποιοι Ευρωπαίοι συνάδελφοι δεν ήταν διατεθειμένοι να παίξουν στεναρό ρόλο. Και αυτό ήταν πολύ λυπηρό. Λέτε ότι χρειαζόμαστε αρκετά κονδύλια που θα δεσμευτούν για αυτό το σκοπό θα πρέπει το ποσοστό του αμυντικού προϋπολογισμού της Συμμαχίας, τον οποίον φέρουν οι ευρωπαϊκές χώρες και ο Καναδάς, το 2007 ήταν περίπου το 32% του προϋπολογισμού της ε, Συμμαχίας και το 12 έπεσε στο 28% του ε, προϋπολογισμού της ε, Συμμαχίας. Κατά αναλογία οι Ευρωπαίοι λοιπόν θέλουν να κάνουν λιγότερα πράγματα και δεν αναλαμβάνουν ευθύνες ε, στον τομέα της άμυνας. Τώρα για την παραγωγή, έρευνα και ανάπτυξη, αμυντικές βιομηχανίες, αυτές κυριαρχούνται από 5-6 χώρες, για να μην πω 2-3 που είναι επικεφαλής στην έρευνα και την ανάπτυξη. Σας παραπέμπω σε μια εξαιρετική εργασία από το Think Tank New Direction που λέγεται White Elephants ε, τα προγράμματα συνεργασίας για την άμυνα στην Ευρώπη που ξεκάθαρα λέγουν ότι δεν χρειάζεται εμπλοκή των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων, θεσμικών οργάνων, ώστε να βελτιωθεί η αμυντική συνεργασία. Δέχεστε ότι τις απόψεις σας θα πρέπει να τις δείτε στο πλαίσιο του νέου ενθουσιασμού που φαίνεται να έχει εκδηλωθεί και μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων υπέρ των ε, διατλαντικών σχέσεων και μάλιστα ο κύριος Λίσεκ σήμερα το πρωί ε, αναφέρθηκε στο Ευρωπαϊκό Εμπορικό Επιμελητήριο που συζητήσαμε αυτά τα θέματα και αντί να φτιάξουμε την Ευρώπη ε, Ω ανταγωνιστή των ΗΠΑ, δεν κινούμεθα προ μια κατεύθυνση όπου θέλουμε η ΗΠΑ να είναι ο προτιμόμενος εταίρος μας. Τέλος, δεν πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αντλήσει διδάγματα και να αρχίσει να, σταματά αυτή την προσπάθεια να αποκτά ε, όλο και περισσότερες αρμοδιότητες. Ήδη έχει πάρα πολλές. Και ένα πολύ καλό παράδειγμα σχετικό και με τη συζήτηση είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος, ο οποίος δουλεύει εξαιρετικά. Υπάρχουν 20 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ε, ανήκουν στον οργανισμό. Δεν είναι δηλαδή ε, ε, οργανισμός της Ευρωπαϊκής, θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να απορροφήσει τον οργανισμό του διαστήματος και ευλόγως κάποια κράτη-μέλη ανθίστανται. Δεν πιστεύετε λοιπόν ότι κινείται την όλη συζήτηση προς λάθος κατεύθυνση. Δεν θα ήταν καλύτερα να δείξουμε εμπιστοσύνη στην ε, συμμαχία, την Ατλαντική Συμμαχία και επειδή έχουμε ε, στιβαρή συνεργασία και καλούς εταίρους όπως ε, είπα θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε προς τα εκεί και να μην αφήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βάλει την γραφειοκρατική της φραγίδα σε εξελίξεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα και εγώ χαιρετήσω τον Επίτροπο με την παρουσία του και παρά τις προηγούμενες του. Νομίζω ότι σημαντικό είναι να υπογραμμίσουμε ότι ήταν και ένας από τους πολύ σημαντικούς ευρωβουλευτές στο παρελθόν. Η παρουσία σας εδώ σήμερα γίνεται στην κατάλληλη στιγμή, διότι χθε κάναμε την ε, συζήτηση που αφορά την εκτίμηση εξωτερικής υπηρεσίας της και νομίζω ότι αποφασίσαμε ότι υπάρχουν και κάποια σαν σε επίπεδο ε, και άμυνας. Είπε κάποιος υπουργός ότι σήμερα έχουμε στρατούς που δεν έχουν αν θέλετε, συμβατικούς εμφανούς εχθρούς, αλλά έχουμε εχθρούς που δεν έχουν ε, ίσως ε, αντικείμενα. Θα πρέπει λοιπόν να πω κύριε Επίτροπε, ότι επί αυτού του θέματο είναι σημαντική η δημιουργία αυτής τη Task Force. Θα ήθελα να κάνω τρεις σημαντικέ και συγκεκριμένε ερωτήσει σε σχέση με αυτό που και ο κύριος Γκάλερ, που ανέφερε τι οδηγίες που εγκρίναμε το 2009. Πόσο κατάλαβα από την παρέμβασή σα, η θέση σε και η εφαρμογή αυτών των οδηγιών δεν δημιούργησε πρόβλημα στα κράτη-μέλη και ο απολογισμό ξέρω ότι θα πρέπει να γίνει το 2017 στο Ευρωπαϊκό Κοινό. Ποια είναι όμω η δική σα εκτίμηση όσον αφορά την ε, ε, θέση εφαρμογή αυτών των οδηγιών. Νομίζω επίσης ότι τα πλαίσια των ε, δυνατοτήτων που έχουμε στην, ε, όσον αφορά τις ένοπλες δυνάμεις Έχουμε ε, μεγάλες δυνατότητες, αλλά στα πλαίσια της ιστορικής υπηρεσίας μπορούμε να κινητοποιήσουμε μόνο γύρω στους πέντε στρατιώτες. Ο κύριος Βανόρντεν επίσης αναφέρθηκε στις δαπάνες σε θέματα άμυνας. Όταν ζητούμε από τους πολίτες της Ευρώπης να μας πούν εάν θα ήθελαν η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει πολιτική, οικονομική και Ευρωπαϊκή Ένωση της Άμυνας, πρέπει να πω ότι γενικότερα παίρνουμε θετικές απαντήσεις. Όταν λέμε όμως ότι θα πρέπει να βάλεις πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτή την πολιτική άμυνα, υπάρχουν ενδιασμοί και βλέπουμε να μειώνονται οι δαπάνες προβλέπονται από τους, στους προπολισμούς. Και τώρα μιλούμε για εξαγωγέ της αμυντικής μας βιομηχανίας σε αναδυόμενες οικονομίες. Αυτό θα ήταν ίσως ε, μία, ένα, μία διέξοδος για τη αμυντική μας βιομηχανία, αλλά έχει και πολλούς περιορισμούς. Εάν δεν μπορέσουμε λοιπόν να κάνουμε μία πραγματική αμυντική βιομηχανία καινοτόμο και ανταγωνιστική, θα χάσουμε το τρέν της τεχνολογίας. Συγκεκριμένη με ερώτηση είναι, σε ποιο μέτρο είναι συμβατές η ατζέντα για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα με της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τους στόχους του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Επίσης, κύριε Επίτροπε, Εκ μέρους της Επιτροπής καταλήξατε σε σαφή συμπεράσματα μετά από τις κρίσεις στην ε, Λιβύη και στο Μάλι για την ε, έλλειψη ε, Monsieur le Vice-président Lisek. Συμβατότητα μεταξύ των διαφορών πλήμων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λίσεκ. Ponieważ parlament jest wielokulturowy i wielojęzyczny, to będę mówił po polsku. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω στα πολωνικά. Ε, έτσι θα ακούσουμε σχεδόν όλες τις γλώσσες που υπάρχουν στην Επιτροπή. Κύριε Επίτροπε, η Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία είναι εν μέρει ανταγωνιστική, εν μέρει όμως δεν είναι, γιατί από τεχνολογικής άποψης δεν είναι η πλέον προηγμένη βιομηχανία και είναι και διάσπαρτη. Έχουμε πάνω από 20 ναυπηγεία που κατασκευάζουν ε, σκάφη, ή είπα έχουν μόνο τρία. Εμείς στην Ευρώπη προσπαθούμε να κατασκευάσουμε ε, στρατιωτικά αεροπλάνα και ε, να παράσχουμε εκπαίδευση. Οι Αμερικανοί έχουν δύο τέτοιες επιχειρήσεις, δύο τέτοιες εταιρείες. Έτσι λοιπόν ε, στην Ευρώπη η ανταγωνιστικότητα μειώνεται γιατί μειώνονται και οι αμυντικοί προϋπολογισμοί. Προφανώς η ζήτηση για στρατιωτικό εξοπλισμό αυξάνεται, αλλά πρέπει να είναι υψηλής τεχνολογίας, ηλεκτρονικοί εξοπλισμοί, όπως μη επανδρομένα αεροσκάφη, αλλά υπάρχει όλο και λιγότερη ζήτηση για τεθωρακισμένα ή άλλα πιο συνήθη ε, πιο συνήθι στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Αυτό επηρεάζει τις αμυντικές βιομηχανίες στα κράτη-μέλη. Θα υπάρξουν και κοινωνικές επιπτώσεις από όλα αυτά που αφορούν την απασχόληση. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξής. Σε αυτήν την ειδική ομάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναλύσατε και μέσα από αυτή την προοπτική το πρόβλημα και βλέπετε κάποια λύση για το μέλλον τι πρέπει να γίνει δηλαδή στην αμυντική βιομηχανία στην Ευρώπη που δεν είναι τόσο αποδοτική, αποτελεσματική, διάσπαρτη, με μικρότερη ζήτηση από τα κράτη-μέλη και ε, με ε, όρια σε σχέση με την ε, εκμετάλλευση που μπορούμε να κάνουμε. Το πρόβλημα είναι σοβαρό νομίζω. Κύριε Ζέμκε. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που και εγώ μπορώ να μιλήσω στα πολωνικά. Να ρωτήσω τον Επίτροπο. Όποτε μιλάμε για κοινή πολιτική άμυνας, ε, παγιδευόμεθα γιατί οι Ευρωπαίοι ηγέτες μιλούν για την ανάγκη εφαρμογής αυτής της πολιτικής για διάφορους λόγους. Ε, η κρίση είναι ένα από τα προβλήματά μας. Έχουμε περικοπή των προϋπολογισμών και όπως είπε και ο προηγούμενος ομιλητής, πολλά έργα, προγράμματα μειώνονται. Το πρόβλημα είναι ότι όποτε εξετάζουμε τα δεδομένα, που είναι και ζωφερά και δεν πρόκειται βραχυπρόθεσμα να αλλάξουν, διαπιστώνουμε ότι δεν μπορούμε σε στρατιωτικό επίπεδο δεν μπορούμε να ε, έχουμε στρατιωτική επιχείρηση για την οποία θα είμαστε υπεύθυνοι εκτός Ευρώπης. Ίσως θα πρέπει να ε, Πρέπει λοιπόν να αξιοποιούμε καλύτερα τα διαθέσιμα κονδύλια για να μην μιλήσω για κοινωτικοποίηση της πολιτικής. Ε, ίσως θα έπρεπε να δούμε πώς μπορούμε να αναλάβουμε μια στρατιωτική επιχείρηση κάπου. Θα πρέπει να είμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε ένα project στην Ευρώπη. Ε, για παράδειγμα αυτά τα καταδιοκτικά γιατί αυτά θα βοηθήσουν ε, σε περίπτωση επιχειρήσεων εκτός συνόρων στην Ευρώπη. Υπάρχει μεγάλη ε, διαφορά και αντίφαση μεταξύ αυτών που κάνουμε και αυτών που λέμε. Ας αλλάξει λοιπόν αυτή η πραγματικότητα και ας βγάζουμε λιγότερους ε, λόγους. Κύριε Επίτροπε, ε, μιλήσατε για την ανάγκη μιας ε, κοινή στόχευσης. Ε, πιστεύω ότι θα πρέπει αυτό να είναι μέλημα των κρατών μελών, των κυβερνήσεων του ΝΑΤΟΥ. Μείνετε έξω από την άμυνα. Αυτό είναι θέμα κρίσιμο για τις εθνικές κυβερνήσεις, ο τομέας της άμυνας. Είδαμε στο, Άμιλ, στο Μάλι ότι οι Γάλλοι τα πήγαν πάρα πολύ καλά, σχεδόν μόνοι και μια μικρή βοήθεια από τους Βρετανούς μεταφορές. Ε, στη Λιβύη επίσης γαλλική επιχείρηση με λίγη αμερικανική υποστήριξη. Ε, νομίζω λοιπόν ότι αυτό σημαίνει σαφές όραμα. Τώρα, για τα συγκεκριμένα ερωτήματα. Αν ε, επικεντρωθείτε στη βιομηχανική πολιτική που ελπίζω να μην είναι τόσο σοβιετική και επικεντρωθείτε στις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις δεν θα περιορίσετε την δυνατότητα ευρωπαϊκών επιχειρήσεων να συνεργάζονται στενά με τη ΣΥΠΑ. Δηλαδή θα αποκλείσετε την ε, κοινή τεχνολογία ε, στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Δεν θα υπονομευόταν έτσι το ΝΑΤΟ. Τέλος, ε, οι συγχωνεύσεις ενδεχομένως έχουν υπονομεύσει την δυνατότητα πολιτικής. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Νομίζω ότι μία από τις πολλά υποσχόμενες εξελίξεις σχετικά με την έρευνα και την ε, καινοτομία είναι η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Συνεργασίας. Είναι κάτι το οποίο επιτρέπει να υπάρξει στενότερη συνεργασία ανάμεσα στην Επιτροπή και τις Ευρωπαϊκές Αμυντικές Βιομηχανίες. Πώς βλέπετε εσείς ε, το θέμα της ε, ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στο νέο αυτό πλαίσιο. Τι μπορούμε να κάνουμε στον τομέα αυτό. Είδα ότι οι δαπάνες για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ε, περιέργως από μία άποψη, κατεξαίρεση αν θέλετε, έχουν αυξηθεί. Τι πιστεύετε ότι ε, μπορεί να προσφέρει το ευρωπαϊκό πλαίσιο συνεργασίας στο θέμα της ασφάλειας των χώρων. Κοιτάξτε, θεωρητικά κύριε Επίτροπε, τώρα έπρεπε να φύγετε, αλλά ε, κοιτάξτε, τελευταίος ο κύριος Γιάννης, ε, τελευταίος σύντομα. Είχα ζητήσει αρκετή ώρα. Δεν ήξερα ότι θα μου δίνατε, εν πάση περιπτώσει, τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον κύριο Μπαριέ για την ομιλία του. και με, το θέμα και με τον κύριο Ταβιάννη έχουν αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το θέμα της κοινοτικοποίηση της βιομηχανίας, ιδιαίτερα στον τομέα της βιομηχανίας της άμυνας. Είναι ένα πρώτο μεγάλο βήμα είναι κάτι που θα συνεισφέρει στην ενότητα της Ευρώπης πέρα από την Ευρώπη και μετά από την Ευρώπη των αγορών, μετά από την νομισματική Ευρώπη, μετά από την κρίση θα υπάρξει μια ένωση πολιτική και οικονομική και μια μεγάλη ανάγκη απέτηση αν θέλετε να υπάρξει και μια ισχυρή πολιτική στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας που δεν είναι ανταγωνιστική με τον ΝΑΤΟ αλλά συνεργάζεται με τον ΝΑΤΟ και δεν είναι ανταγωνιστική αλλά συνεργάζεται και με τα Ηνωμένε Πολιτείε. Άλλωστε και ο ίδιος ο πρόεδρος Ομπάμα σημείωσε το ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών για μια ισχυρότατη Ευρωπαϊκή Ένωση ιδιαίτερα στον τομέα αυτό της ασφάλειας και της άμυνας. Και αναφέρομαι εδώ στην παρέμβαση της Γαλλίας στο Μαλί, και που δεν θα μπορούσε ίσως να έχει συμβεί αν δεν υπήρχε μια στήριξη ευρωπαϊκή. Παραδόξως λοιπόν η κρίση και η δημοσιονομική δυσφορία βοηθά προς την κατεύθυνση αυτή. όχι με μικρότερους προϋπολογισμούς, αλλά με τους ίδιους προϋπολογισμούς σωστότερα χρησιμοποιημένους και αυτό συμβαίνει ακριβώς και με την ε, βιομηχανία, ε, την πολεμική βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είπαν και οι συνάδελφοι θα πρέπει να υπάρξει ενοποίηση των προσπαθειών. Είναι πάρα πολύ προφανές αλλά και δύσκολο να προχωρήσουμε, είναι δύσκολο να πείσουμε τους σκεπτικιστές, αλλά ελπίζω ότι με τον κύριο Μπαρνιέ οδεύουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα απαντήσω επιγραμματικά. Σημείωσα με μεγάλη προσοχή τις ε, υποδείξεις σας, τις ερωτήσεις που μου κάνετε και θα συνεχίσουμε φαντάζομαι το διάλογο δεδομένου ότι ε, η εργασία που τελειούμε είναι εργασία που θα διαρκέσει στο χρόνο. Τώρα, οι δύο τελευταίες ε, παρεμβάσεις είχαν διαφορετικό περιεχόμενο του κυρίου Γιάννη και του κυρίου Βλέπουμε ότι μεταξύ των δύο πεπιθήσεων που εκφράσατε, τις οποίες σέβομαι, αν και είμαι πιο κοντά στη μία ε, παρά την άλλη, πρέπει να βρούμε τη μέση εδώ, Τη χρυσή τομή. Πιστεύω ότι γενικά για την αμυντική βιομηχανία υπάρχουν πολλοί λόγοι και υποχρεώσεις δεδομένης της ε, συγκύριας και το πόσο μας ενδιαφέρουν τα θέματα της ασφάλειας και της άμυνας, ώστε να θέσουμε από κοινού τα μέσα που διαθέσουμε. Ακόμη και σε επίπεδο Βρετανικής αμυντικής βιομηχανίας ε, η ανάγκη αυτή εκφράζεται. Όταν δούμε ποια είναι η διμερής ε, συμφωνία η οποία έκανε η Γαλλία με την Αγγλία. Παρά το γεγονό ότι δεν μπορούμε να συνοψίσουμε όλοι μα την ευρωπαϊκή πολιτική σε αυτή τη διμερή συμφωνία, σε αυτή όμω τη διμερή συμφωνία έχουμε την απόδειξη ότι Γάλλοι και Βρετανοί έχουν ανάγκη να συνεργαστούν για να ενισχυθούν αμοιβαίω. Πιστεύω λοιπόν και εγώ, όπως πολλοί από εσά, ότι αυτό δεν ισχύει μόνο για τους ε, εξοπλισμούς ή για την ασφάλεια της Γαλλίας, της Βρετανίας, είναι κάτι το οποίο ισχύει για τις 27 χώρες μέλη, που έχουν κατά το μάλλον ήτον στρατηγικά και στρατηγικά παρεμφερή ενδιαφέροντα. Και πιστεύω ότι αν ο καθένας παραμείνει μόνος του για να ενεργήσει, θα είναι πιο αδύναμος. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε την κοινή την ενιαία αγορά της βιομηχανίας γενικότερα και της αμυντικής βιομηχανίας ειδικά και για να είμαστε και αυτό για να μπορέσουμε να είμαστε και πιο ισχυροί και πιο αποτελεσματικοί στις εξαγωγές. Τηλεγραφικά. Θα πω τώρα στον κύριο Κάλαμ ότι όντως ε, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι ένα από τα κύρια θέματα που μας απασχολούν. Αυτό είναι ε, κάτι το οποίο συζητήθηκε και η κυρία Κρόης το ανέφερε και στην διάσκεψη που είχαμε στο Μόναχο. Όντως το θέμα αυτό είναι ένα από τα θέματα με τα οποία ασχολείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το θέτει επιτάπητος και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο προς συζήτηση. Κύριε Γιάννη. Ξέρουμε ότι σήμερα δεν έχουμε περισσότερους πόρους οικονομικούς, ούτε θα έχουμε περισσότερο στο μέλλον, άρα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους διαθέσιμους πόρους και είμαι πεπισμένος ότι πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε τα κοινοτικά κονδύλια καλύτερα. Δηλαδή να κάνουμε κοινά προγράμματα ε, για θέματα στρατηγικής σημασίας, το τομέα αυτό που μας ενδιαφέρουν και τα χρησιμοποιήσουμε καλύτερα να είμαστε πιο αποδηματικοί. Επίσης υπάρχει το θέμα της, ρυθμι... της ε, κανονιστικής αρμοδιότητας που έχουμε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο με την ε, εμπειρία που έχουμε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε επωφελώς. Στο μη στρατιωτικό τομέα το έχουμε χρησιμοποιήσει, ανέφερα, και πολλούς τομείς στους οποίους στα πλαίσια της ε, εντολής που έχουμε δώσει μπορούμε να προχωρήσουμε για κοινού κανόνες, για προδιαγραφές σε διάφορους τομείς. Μίλησα εγώ για την ε, αεροπλοή, για τις αεροπορικές μεταφορές και τις δυνατότητες που έχουμε και την εμπειρία, την πραγματομοσύνη, την χρησιμοποιούμε σωστά. Νομίζω ότι θα πρέπει ό,τι διαθέτουμε σε αυτό το τομέα να το χρησιμοποιήσουμε καλύτερα. Επίσης, αυτό το οποίο μας απασχολεί κυρίως και εγώ γενικότερα μίλησα για τη βιομηχανική πολιτική και ειδικά για την αμυντική ε, βιομηχανία είναι η βούληση σε κάθε μία από τις χώρες μας όπου υπάρχει να συνεχίσει να υπάρχει και να παγιωθεί η δυνατότητα παραγωγής στην Ευρώπη. Και να διατηρήσουμε τις τεχνολογίες μας και τις ικανότητες που έχουμε στον τομέα της αβιοντιμητικής μας βιομηχανίας. Και αυτό πολλές φορές είναι ένα θέμα ε, το οποίο δημιουργεί ερωτηματικά. Γι' αυτό σας είπα τι ακριβώς κάνουμε εμείς για να βοηθήσουμε τα κρατημέλη από τη μεριά της Επιτροπής. Ο κύριος Αλαφράνκα η κυρία Νίτς, ο κύριος Γκάλερ ανέφεραν τα θέματα του προπολογισμού, ο κύριος και επίσης. Και όπως είπε και η κυρία Νέτ, θα πω και εγώ ότι έχουμε, βλέπουμε να μας ενείται ένα νέο παράθυρο δυνατοτήτων, ευκαιριών. Ναι, άνοιξε το παράθυρο, όχι μόνο για θέματα τα οποία αφορούν μόνο τον προπολογισμό, ο οποίος μειώνεται, αλλά σε σχέση και με τις νέες απειλές. Και τελικά, σε σχέση με τις νέες στρατηγικές επιλογές των ΗΠΑ. Γι' αυτό για αυτούς του τρεις λόγους υπάρχει αυτό το παράθυρο, άνοιξε, θα μπορέσουμε να δράξουμε αυτή την ευκαιρία. Δεν έχω απάντηση. Μπορείτε ε, επί αυτού του θέματος να κάνετε και διάφορες ερωτήσεις στην κυρία Άστον και στι κυβερνήσει σας. Εγώ δεν χρειάζεται να μου υπενθυμίσει κανείς ότι η αρμοδιότητα σε θέματα ασφάλειας και άμυνας είναι κατά πρώτον και πρώτη στο λόγο στα χέρια των κρατών μελών. Αλλά Ξέρουμε ότι υπάρχει και αυτό ο ειδικό σύνδεσμος που έχει δημιουργηθεί και θα πρέπει να τον χρησιμοποιήσουμε. Είμαι πεπισμένο ότι αυτές τις νέες λοιπόν θα δράξουμε εάν τα προγράμματα και τους πόρους τους χρησιμοποιήσουμε προς κοινό όφελος και κάνουμε μία σωστή στρατηγική. Και το ερώτημα που θα θέσουμε στα κράτη-μέλη, θα μπορούσαμε στην λευκή μας βίβλο να θέσουμε, όπως αναφέρεται, είναι Ποια είναι η αμυντική, ε, με συγχωρείτε, η βιομηχανική βάση που διαθέτει η Ευρώπη για να αντιμετωπίσει αυτές τις απειλές, ποιες είναι οι, ποιοι είναι οι πόροι που μπορούμε να κινητοποιήσουμε για να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση. Και βεβαίως, χωρίς να ξεχνούμε το θέμα της ανεξαρτησίας, της αυτονομίας της Ευρώπης. Βεβαίως, ε, πρέπει να σας πω ότι εγώ είμαι υπέρμαχος της ε, διατλαντικής ε, συμμαχίας και συνεργασίας. Βεβαίως θα πρέπει ότι γίνει να γίνει η όρης, ώστε να είμαστε και εμείς αξιόπιστοι. Το είπαν οι Αμερικανοί. Για να είστε αξιόπιστοι πρέπει να υπομειστείτε τις ευθύνες σας. Και είμαι υπέρ της διετής και ενίσχυσης του ΝΑΤΟ. Είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ, μέλη της συμμαχίας, αλλά ενθυμίστε ότι υπάρχει ένα έγγραφο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, το έγγραφο το περίφημο του Σαμαλό, όπως λέγεται, μεταξύ Γάλλων και Βρετανών, αυτόνομη και αλληλέγγυη ε, συνεργασία και συμμαχία. Μιλήσατε για τον Άτο Κοινωνόδο. Ξέρετε πολύ καλά, τέλος πάντων, εγώ ξεπερνάω λίγο τα όρια του Επιτρόπου γιατί είμαι και πολιτικός. Ξέρετε ότι υπάρχουν επιχειρήσεις και κρίσεις στις οποίες δεν θέλει να δεσμευσει τον, ε, το ΝΑΤΟ. Αναφέρω την κρίση, το πρόβλημα του Μαλή δεν μπορεί να αναλάβει δεσμεύσεις. Τη γεωργία σας υπενθυμίζω. Άρα η πολιτική ασφάλειας, η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας μας δίνει και μια ευελιξία ακόμη και για να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε με ευφύ τρόπο και συνεργαζόμενοι τους Αμερικανούς για να ανταποκριθούμε σε αποκλήσεις ε, στρατιωτικού και μη στρατιωτικού χαρακτήρα που εμφανίζονται ανά τον κόσμο και οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ίσως για να απαντήσω και στον κύριο Γκάλερ θα πω ότι δεν έχω πρόβλημα, μπορούμε να συμμετάσχουμε όλοι για τη δημόρφωση της Λευκής Βίβλου. Η κυρία Νέτς και ο κύριος Γκάλερ μου είπαν ποια είναι η άποψη των κρατών μελών όσον αφορά τις εργασίες που αναλάβει Task Force. Μετά από πρόσκληση της κυρίας Άστον, παρουσίαση υπουργού Άμυνα στην ε, τελευταία συνεδρίασή του το όλο θέμα της Task Force και πρέπει να πω ότι η πρωτοβουλία αυτή έτυχε υποστήριξη διότι πιστεύουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και οι 27 κυβερνήσεις ότι υπάρχει μία προστιθέμενη αξία με την δουλειά που επιτελείται και πρέπει να συνεχιστεί. Κύριε Γκάλερ, μου κάνετε κάποια δύσκολα ερωτήματα. Δεν έχω απάντηση. Αν χρειάζονται δύο διαφορετικές υπηρεσίες μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και της Επιτροπής, και αν δεν θα πρέπει αυτός ο οργανισμός να χρηματοδοτείται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας συμμετέχει στις εργασίες της Task Force. Διαφορετικά δεν θα είμαστε σωστοί και έξυπνοι. Τώρα, όσον αφορά τη χρηματοδότηση όλων αυτών των προγραμμάτων και μέσων, νομίζω θα πρέπει να είμαστε πραγματιστές. και να μην προσπαθούμε να κινήσουμε τα πάντα για να βρούμε πόρους από παντού. Τώρα, πριν από το εαρινό, ε, συγγνώμη, πριν από το καλοκαιρινό, πριν από ε, την διάσκεψη, τη θερινή διάσκεψη κορυφής, νομίζω ότι έχουμε μήνες μπροστά μας για να προετοιμαστούμε κατάλληλα για να παρουσιάσουμε καλύτερα τα θέματα που θα έχουν σχέση με την αποδοτικότητα και την θέση από κοινού των μέσων που διαθέτουμε. Αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή ασχολούμεθα με τις δύο ειδικέ οδηγίες για τις ε, κρατικές προμήθειες, δημόσιες συμβάσεις και την ε, αδιαδότηση. Από πέρσι το καλοκαίρι άλλαξαν πολύ τα πράγματα με θετικό τρόπο, κυρίως για την μεταφορά των ε, δημοσίων συμβάσεων. Μία χώρα μόνο ακόμη, το Βέλγιο, δεν έχει μεταφέρει στο εθνικό του δίκαιο την οδηγία αυτή, αλλά βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης και το θέμα των παραβιάσεων επίσης, καθώς και τα εκτελεστικά ε, θα ε, περατωθεί. Ακόμη τα εκτελεστικά μέτρα δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή από όλες τις χώρες, αλλά θα ολοκληρωθούν επίσης σύντομα. Όσον αφορά για την οδηγία για τις ε, κρατικές προμήθειες, γιατί άλλες είναι θέμα ευθύνης του κυρίου Ταγιάννη, η τελευταία χώρα που δεν είχε ολοκληρώσει την μεταφορά στο εθνικό δίκαιο ήταν η Ολλανδία, αλλά ε, αυτή την εβδομάδα ολοκλήρωσε το όλο θέμα. Τώρα, υπάρχουν ακόμη τεχνικές λεπτομέρειες που πρέπει να επεξεργαστούμε ακόμη. Επίσης, θα ήθελα να πω στον κύριο Σοφοκλέους, όπως είπα και στον κύριο Ζέμ και στον κύριο Λίζεκ, ότι χρειαζόμαστε για να διευκολύνουμε όλες αυτές τις τεχνικές αποφάσεις και πολλές φορές οικονομικές ή νομικού χαρακτήρα, να συμφωνήσουμε σε μία στρατηγική και αυτή την στρατηγική για την αγορά της αμυντικής βιομηχανίας ε, μελετούμε και επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Ακούγοντα τον κύριο Βανόρντεν προηγουμένω, που πάντα ε, είναι πάρα πολύ ευθύ αυτά που ζητά, αλλά και εγώ το ίδιο κάνω, σκέφτηκα κάτι που άκουσα τώρα τελευταία, που είναι αυτά τα οποία είπε ο κύριος Άστον Κάρτερ στο Μόναχο, ε, αναπληρωτής υπουργός άμυνας τον είπα. Θα πρέπει δηλαδή να ακούσετε τι είπε για να δείτε πώς οι Αμερικανοί που είναι οι κύριοι εταίροι μας αντιλαμβάνονται την άμυο. Ο κύριος Κάρτερ πέντε φορά στην ομιλία του μίλησε για προστασία των ε, Αμερικανικών αμυντικών βιομηχανιών. Και ακούγοντάς τον είπα, όντας εγώ υπέρμαχος της ε, διατλαντικής συνεργασίας και πρέπει να πω ότι προσπάθησα στην Ουάσιγκτον να συζητήσω όλα αυτά τα θέματα και στα πλαίσια εταιρικών σχέσεων σε εμπορικό επίπεδο που είσαι και ο πρόεδρος Ομπάνα, είπα ότι όσον αφορά την αμυντική βιομηχανία, ότι αυτό που δεν μπορούν αν δεν κάνουν κάτι Ευρωπαίοι για τον εαυτό τους, να το κάνει κανένας για πάρτι τους. Εμείς λοιπόν, οι ίδιοι και για μας τους ίδιους πρέπει να κάνουμε πράγματα τα οποία κανένας δεν θα τα κάνει, αν τα κάνουμε εμείς. Γι' αυτό επειδή πιστεύει ότι μπορεί να είναι χρήσιμη η Επιτροπή, σύστησε αυτή την Task Force και βεβαίω, όπως είπατε κύριε Πρόεδρε θα προσπαθήσω ώστε να ενημερώνεστε στο Κοινοβούλιο για το τι γίνεται και τους επόμενους μήνες θα έχετε περισσότερα νέα από τον τρόπο λειτουργίας Task Force. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Συγγνώμη που σας καθυστερήσαμε λίγο περισσότερο από ό,τι είχε προβλεφθεί, αλλά νομίζω ότι άξιζε τον κόπο. Και αφού ακούσουμε και τον κύριο Ταγιάννη, σε μερικού μήνε ελπίζω θα μπορέσουμε να έχουμε το φθινόπωρο μια κοινή συνεδρίαση με εσά τους δύο για να κάνουμε απολογισμό τη όλης κατάσταση πριν από το Συμβούλιο του επομένου Δεκεμβρίου. S'il Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ. Θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Καλωσορίζουμε τον κύριο Ποπόφσκι, αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα της ε, Εξωτερικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μαζί του θα αναφερθούμε στο άτυπη συνάντηση των Υπουργών Άμυνα που έλαβε πριν μια εβδομάδα χώρα στο Δουβλίνο. Πρόκειται για ένα από τα πρώτα βήματα προς την προετοιμασία του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου που θα συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων και την κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας. Και βεβαίως ε, στην συνάντηση αυτή μελετήθηκαν και άλλα θέματα επικαιρότητα. Το, η κατάσταση στο Μαλί. Ε, ξέρουμε ότι επισήμω ε, τέθηκε σε εκκίνηση και η νέα αποστολή UETM στο Μαλί. Υπάρχουν ακόμη, όπως ξέρουμε, σε συγκεκριμένα στιγμή κάποια ερωτηματικά, κάποια κενά, θα μας ενημερώσετε. Και Ξέρουμε ότι συζητήθηκαν και θέματα που αφορούν άλλες αποστολές και ξέρω ότι εχθές έπρεπε να δούμε και πώς θα κάνουμε τον ορισμό αυτού της διαχείρισης κρίσεως για το πρόβλημα της Λιβύης. Γίνεται λόγος για αυτό το θέμα εδώ και ένα χρόνο συγκεκριμένα. Φορτωμένη λοιπόν η μερίσια διάταξη που είχατε. Και βεβαίως εκ μέρους των ε, συναδέλφων, πρέπει να σας πω πολλών συναδέλφων, ε, μας απογοήτευσε το ότι δεν μπορούσε να προεδρεύσει του συμβολίου αυτού του άτυπου η κυρία Άστον, διότι βεβαίως ήταν για σοβαρούς λόγους, διότι παρέστη του Συμβουλίου Ασφαλείας, συνάντηση που έχει τον ΟΗΕ στην Νέα Υόρκη, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να πω ότι εμένα με ενοχλεί κάπως που για κάποιες προγραμματισμένες τέτοιου είδους συναντήσεις που γίνονται σε τακτά διαστήματα για τόσο σημαντικά θέματα όπως η άμυνα δεν μπορεί να παραστεί είπατε εκπρόσωπος. Όπως είπατε, περίπου η μισή Υπουργή ήταν παρόντα στο Δουβλίνο. Ενώ λοιπόν λέμε ότι το 2013 πρέπει να είναι έτος με μεγάλη σημασία στην ΚΕΠΑ και για να επαναλάβω αυτά τα οποία είπε ο Επίτροπος Μπαρνιέ, θα πω ότι η, πολιτική άμυνας είναι κάτι το οποίο είναι θέμα ευθύνης από ό,τι ισχυρίζονται τα κρατη αλλά θα πρέπει να απομιστούν και την ευθύνη αυτή. Εάν λοιπόν σε μια τέτοια συνάντηση δεν ήταν ούτε καν η μισή Υπουργή Άμυνας, με πραγματικά ποιες είναι οι προτεραιότητες για τα κράτη-μέλη και πώς ιεραρχούνται. Τέλος πάντων, μετά από αυτή την επικριτική παρατήρηση, με μεγάλη ευχαρίστηση σας δίνω το λόγο για να ακούσουμε τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε αυτό το άτυπο συμβούλιο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο πράγματα θα κάνω. Καταρχήν θα αναφερθώ στις συζητήσεις στο Δουβλίνο και μετά θα αναφερθώ και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αν μου επιτρέπετε. Η προετοιμασία της συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ήταν το πιο σημαντικό θέμα μας. Ο Ιρλανδός πρόεδρος Σάκερ ήταν ο πρόεδρος ε, εξ ονόματος της κυρίας Άστον που ήταν στη Νέα Υόρκη και στην Ουάσιγκτον. Ήταν μία συνάντηση ε, που είχε πρωτιά για πολλά θέματα. Πρώτη φορά μιλήσαμε ε, για την άμυνα, δεύτερον ε, πρώτη φορά έγινε στην Ιρλανδία μαζί με τον επικεφαλής των ειρηνευτικών δυνάμεων. Πρώτη φορά ήταν ήταν και ο επικεφαλής στρατηγός για το Μάλι, ο επικεφαλής στρατηγός για τη Σομαλία και ο Ναύαρχος ε, ε, υπεύθυνο για το πρόγραμμα Ταλάντι. Επίσης, ε, πρώτη φορά στο Συμβούλιο έγινε επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ στην Ιρλανδία και για τους οικοδεσπότες ήταν σημαντική εκδήλωση γιατί εκεί οι οικοδεσπότες μας επιβεβαίωσαν τη συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο για κοινή ανάπτυξη ε, εκπαιδευτικών δυνάμεων στο Μάλι, που αυτή είναι μια ιστορική περίσταση και από τη δική τους πλευρά. Λοιπόν, καταρχήν η συζήτηση για την προετοιμασία για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Νομίζω ότι το κλίμα είναι καλό. Υπάρχουν πολλές προσδοκίες, αλλά όλοι θεωρούν ότι αυτή είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Ο Επίτροπος Μπαρνιέ μίλησε για παράθυρο ευκαιρίας που είναι διάπλατα ανοιχτό πρέπει να πούμε και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Η στόχευση της συζήτησης ήταν στις ικανότητες, έγιναν παρουσιάσεις και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα για την Κομισιόν. Δεν θα πω πολλά γιατί τα είπατε με τον κύριο Μπαρνιέ. Παρουσίασε πέντε τομεί ενδιαφέροντα στην εσωτερική αγορά μεγαλύτερες ευκαιρίες αγοράς για τις ε, εταιρείε και τις μικρομεσαίες, τυποποίηση, πιστοποίηση, έρευνα και καινοτομία, ευκαιρίες ε, για έρευνα και ανάπτυξη σε ε, τομείς τεχνολογιών διπλής χρήσης ή σκοπιμότητας, στον κυβερνοχώρο, τεχνολογίες, ε, ε, επιτήρηση εποπτείας στη θάλασσα κλπ. Από τις συζητήσεις ε, τα σημαντικότερα θέματα ήταν τα εξή. Οι περισσότεροι συμφωνούν ότι χρειάζεται στρατηγική αφήγηση από πάνω προς τα κάτω. Οι αρχικοί κρατών και κυβερνήσεων πρέπει να δώσουν κατευθύνσεις προς τα που θα κινηθούμε. Ε, χρειάζεται καθοδήγηση λοιπόν. Ένας υπουργός το παρουσίασε γλαφυρά και είπε η άμυνα έχει σημασία. Αν συμφωνήσουμε όλοι ότι η άμυνα μετράει, πρέπει να συνάγουμε συμπεράσματα και για τις ικανότητες και για τον επενδυτικό μας σχεδιασμό. Πολλοί υποστήριξαν την ανάπτυξη ε, προγραμμάτων σε τεχνολογίες διπλής χρήσης στον κυβερνοχώρο και στο UAS, όπως του λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πολλά κράτη-μέλη υποστηρίζουν ε, περιφερειακές πολυμερείς εισπυρώσεις, ε, δηλαδή το pooling and sharing, αυτή η, κοινή, η συνένωση και η κοινή χρήση ε, και σε περιφερειακό πλαίσιο να γίνεται. Ο ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων υπογραμμίστηκε ιδιαίτερα. Αυτό είναι σημαντικό θέμα για όλους. Και οι μικρότερες χώρες ακόμη που δεν έχουν αξιόλογες αμυντικές βιομηχανίες μπορεί να είναι ε, σημαντικός εταίρος στην αξιακή αλυσίδα της ε, αμυντικής παραγωγής. Ε, μιλήσαμε και για δομές διαχείρισης κρίσεων, αλλά δεν ήταν πολύ σημαντικό θέμα συζήτησης αυτό. Δεν υπήρξαν επίσημα συμπεράσματα, αλλά αν επιχειρήσουμε να συνοψίσουμε τα κύρια θέματα που προέκυψαν από τη συζήτηση, είναι πρώτα απ' όλα ότι είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να δρά, όχι μόνο να είναι πρόθυμη να δρά, θα πρέπει να μπορεί να δρά, να είναι ικανή. Ο εθνικός αμυντικός σχεδιασμός των κρατών μελών πρέπει να μελετηθεί για να δούμε την διασύνδεση, τη σχέση που υπάρχει μεταξύ των σχεδιασμών σε εθνικό επίπεδο και στην ευρωπαϊκή διάσταση. Βεβαίω υπάρχει μια διαδικασία στο ΝΑΤΟ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αξιοποιηθεί δηλαδή και στο ενωσιακό πλαίσιο. Αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε. Και επίσης η συμφωνία για εργασίες σε περιφερειακές εισπυρώσεις. Κλάστερ. Επίσης οι πόροι μετρούν έχουν σημασία. Δεν θα δοθούν περισσότερα κονδύλια για αμυντικούς εξοπλισμούς, αλλά πρέπει να μεγιστοποιήσουμε τις συνέργειες, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη με τα διαθέσιμα κονδύλια, όπως ε, ε, παρουσίασε το θέμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, πάμε στο επιχειρησιακό κομμάτι, το κομμάτι που είναι αφιερωμένο στις επιχειρήσεις. Στο Συμβούλιο Υπουργών, το πρώτο θέμα ήταν το Μάλι. Έγινε μια παρουσίαση από τον ε, Γάλλο Υπουργό για την κατάσταση των πραγμάτων. βεβαίω αλλάζει μέρα τη μέρα η κατάσταση, οπότε δεν θα μπω σε λεπτομέρειες εδώ. Έγινε μια πρώτη παρουσίαση από το διοικητή της αποστολής, τον ε, στρατηγό Λεκουάντ, που έκανε μια ανασκόπηση των προετοιμασιών για την αποστολή και την επιτόπια κατάσταση. Υπάρχουν κίνδυνοι, ε, συμβατικές επιθέσεις δεν είναι τόσο πιθανές στο Μάλι, αλλά μπορεί να υπάρξουν τρομοκρατικά σύμμετρα πλήγματα ε, σε κάποιες περιοχές, γι' αυτό υπάρχει και ανάγκη για κατάλληλη προστασία της αποστολής. Ε, στο φως της κατάστασης των ε, ενόπλων δυνάμεων του Μάλι χωρίς στρατιωτικές υποδομές, το θα πρέπει να υπάρξει μία προσέγγιση συνδυασμένη και για εκπαίδευση, αλλά θα πρέπει να υπάρξει και μια διαδικασία συγκρότησης ε, δυνάμεων ε, στις ένοπλες δυνάμεις. Ο στρατό ε, στο Μαλί χρειάζεται επίσης εξοπλισμούς. Τα κρότη μελη αν επιθυμούν, θα παράσχουν αυτούς τους εξοπλισμούς και εμείς στην εξωτερική δράση θέλουμε να διευκολύνουμε, να παίξουμε ένα ρόλο που θα διευκολύνει τι τις οργανωτικές και την ε, αποστολή που αναπτύσσεται εκεί ε, από την Αφρικανική Ένωση, την αφίσμα. Ε, τρεις πυλώνες θα πρέπει να θεσμοθετηθούν. Τα ελικόπτερα για την εκένωση για ιατρικούς λόγους, τα νοσοκομεία, η ιατρική υποδομή και η προστασία. Θα πρέπει πριν από την αποστολή να υπάρχουν αυτά εμείς ε, είχαμε πρόβλημα με τα ελικόπτερα που δεν ε, υπήρχαν αρκετά, αλλά αυτό το πρόβλημα λύθηκε γιατί έκανε μια προσφορά η βελγική κυβέρνηση που επιβεβαιώθηκε τη Δευτέρα και το Συμβούλιο επήρε την επίσημη απόφαση. Θα υπάρχουν μέχρι τα μέσα Μαρτίου ελικόπτερα διαθέσιμα για την αποστολή και μετά η διαδικασία τέταρτης γενιάς θα ολοκληρωθεί. Τα κράτη-μέλη είναι πρόθυμα να συμβάλλουν, είναι αρκετά καλό το επίπεδο ετοιμότητας. Ε, είχαμε πολλές συνεισφορές και για προστασία. Υπάρχει, ε, ε, ε υπάρχουν 17 περίπου ε, ε, εκπαιδευτές εκεί και θα μπορούσε η εκπαίδευση να αρχίσει αρχές ε, Απριλίου και σας είπα για ένα μηχανισμό ο οποίος δρά διευκολυντικά και υποστηρικτικά. Υπάρχει και μια διάσταση από τα Ηνωμένα Έθνη. Γίνονται συζητήσεις στη Νέα Υόρκη τώρα σχετικά με τον μετασχηματισμό της Αφρικανικής Αποστολής που είναι επιτόπου εκεί και να γίνει η ειρηνευτική αποστολή των Ηνωμένων Εθνών ε, Μπορεί δηλαδή να αναλάβουν οι κιανόκρανοι την ε, αποστολή αυτή. Για να γίνει αυτό όμως θα πρέπει να τροποποιηθεί η νομική βάση και μάλλον χρειάζεται καινούριο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αυτό τώρα το επεξεργάζονται στη Νέα Υόρκη, τώρα που μιλάμε γίνεται αυτό και θα χρειαστούν κάποιες μήνες ούτω ώστε να αλλάξει διεύθυνση η αποστολή και είμαστε σε συνεχή επαφή με το, τα Ηνωμένα Έθνη σχετικά με το τι μπορούμε και εμείς να κάνουμε ούτω ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η ε, αλλαγή. Μια σημαντική διάσταση του EUTM είναι στοχευμένη εκπαίδευση για τους στρατιώτες του Μαλή και για το ανθρωπιστικό δίκαιο και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό το είπαν πολλά κράτη-μέλη. Δηλαδή θα τους εκπαιδεύσουμε στα θέματα αυτά τους στρατιώτες του Μαλή και θα προχωρήσουμε λίγο περισσότερο ε, σε σχέση με το πλαίσιο της αποστολής. Θέλουμε και παρατηρητέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων και από την Αφρικανική Ένωση και από μη κυβερνητικέ οργανώσεις από την Αφρική. Έχουμε διασφαλίσει χρηματοδότηση για το πρόγραμμα αυτό και θα αρχίσει να τρέχει τις επόμενες εβδομάδες. Τώρα, για το κέρας της Αφρικής συζητήθηκε και αυτό και την ε, επιχείρηση Αταλάντη στη Σομαλία ή Αταλάντη είχε μεγάλη επιτυχία. Ιδιαίτερα αν δούμε τα στατιστικά στοιχεία και την ε, ευνίδια μείωση των ε, πειρατικών επιθέσεων τις τελευταίους μήνες, βλέπουμε ότι είναι πολύ σημαντική. Ήταν 176 επιθέσεις το 2011 και μόνο 36 το 2012. Οπότε πάμε σίγουρα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν πρέπει να επαναπαυθούμε, θα πρέπει να συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε. Το, η αποστολή UTM, η αποστολή για την εκπαίδευση για τη Σομαλία θα περάσει από την Ουγγάντα στο Μογκαντήσου, γιατί στην Ουγγάντα λαμβάνει η χώρα τώρα, πάει στο Μογκαντήσου, για αν το επιτρέψουν οι καταστάσεις στον τομέα της ασφάλειας. Δουλεύουμε πάνω σε αυτό τον τομέα. Αυτό θα συμβεί τους επόμενους μήνες. Πέρα από αυτά έγινε συζήτηση για τη συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη ε, αυτό το ΕΦΕ του 2014, απόσυρση από το Αφγανιστάν που θα απελευθερώσει σημαντικούς πόρους στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα μπορούσαν να δοθούν σε ειρηνευτικές αποστολές των Ηνωμένων Εθνών. Είμαστε ο μεγαλύτερος συνεισφέρον στις ειρηνευτικές αποστολέ των Ηνωμένων Εθνών. Λέει, σε ό,τι αφορά τις ε, δυνάμεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λιγότερο από 5% των δυνάμεων. Αυτό μπορεί να αλλάξει. Ε, θα μπορούσε να αλλάξει μετά το 2013. Αυτά ήταν τα βασικά θέματα. Και πολύ σύντομα να προσθέσω κάτι ακόμη. Τη διαδικασία μέχρι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Δεκέμβριο τα συμπεράσματα του περσινού Δεκεμβρίου ε, προσδιορίζουν σαφώς το χρονικό ορίζοντα για τη συζητήση στο CSDP. Τα κράτη-μέλη που θέλουν να, συμβάλλουν, θέλουν να συμβάλλουν, και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί δεν μπορούμε μόνοι μας. Επίσης θα οργανώσουμε έναν αριθμό εκδηλώσεων, σεμιναρίων, διασκέψεων. Για την ίδια τη διαδικασία βλέπουμε την προετοιμασία σε δύο φάσεις. Μια άτυπη μέχρι το Σεπτέμβριο, όπου θα δούμε θέματα και προτεραιότητες θα τα διερευνήσουμε και θα ψάξουμε να δούμε ποια θα είναι τα παραδοτέα ε, από τη συζήτηση αυτή αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων θα δούμε συγκεκριμένα παραδείγματα αμυντικών συνεργασιών και θα αντλήσουμε διδάγματα και από το Μαλί, από το παρελθόν. Από τη Λιβύη θα δούμε τις μάχημες ομάδες που αναφέρθηκαν στη συζήτηση με τον Επίτροπο Μπαρνιέ και πρόθεσή μας είναι να το βάλουμε στην εμερήσια διάταξη των Υπουργών Άμυνα στην επόμενη συνεδρίαση τον Απρίλιο στο Λουξεμβούργο και θα ακολουθήσει μετά μια τυπική επίσημη φάση μετά το καλοκαίρι. Γιατί είπα ότι εκπρόσωπος θα παρουσιάσει μια έκθεση για το αντικείμενο αυτό μέχρι το Σεπτέμβρη. με βάση το προηγούμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και με βάση την εμπειρία από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και τους τον οργανισμό και μετά θα έχει εγκριθεί και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αμυντική βιομηχανία και τις αγορές. Και ε, με, πάνω σε αυτή τη βάση η Προεδρία του Συμβουλίου θα ε, ε, θεσπίσει, θα εκδώσει συστάσεις και τα συμπεράσματα. Τώρα, για τις συσπυρώσεις, τα clusters αυτά, ε, πάνω στα οποία θα εργαστούμε για να παραμείνουμε στοχευμένοι. Θα αξιοποιήσουμε όλες τις ευκαιρίες για, την επι... να υπάρξει πρόοδος. Αναφέρθηκα στο... στο Συμβούλιο του Απριλίου. Το Μάρτιο επίσης ε, είναι ένα σημαντικό ραντεβού με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας που θα συζητηθούν πολλά από αυτά τα θέματα. Έτσι λοιπόν Απαιτείται να μην χάσουμε την ευκαιρία αυτή και να προσπαθήσουμε να ξεφύγουμε λίγο από την πεπατημένη. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία και το Συμβούλιο έχει ήδη ξεκλειδώσει θα έλεγα ορισμένα θέματα. Εφόσον προετοιμαστούμε με σωστό τρόπο αυτό θα φανεί χρήσιμο. Συνδέεται η διαδικασία που οδηγεί στο Συμβούλιο από τη μία και ε, στην επανεξέταση των διαδικασιών γύρω από την Ευρωπαϊκή Εξωτερική Δράση, και την Υπηρεσία Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Δράσης. Αυτά είναι θέματα, θα πρέπει να μας δείξουν τον τρόπο με τον οποίο έχουμε λειτουργήσει μέχρι τότερα, τον τρόπο με τον οποίο έχουμε εργαστεί μέχρι τότερα. Οι συζητήσεις γύρω από τα θέματα αυτά είχαν ήδη ξεκινήσει τον μήνα Σεπτέμβριο. Έχουμε λίγο χρόνο λοιπόν για εφάνταστες αν θέλετε ιδέες. Δεν θα πρέπει να βιαστούμε να καταλήξουμε σε κλειστά συμπεράσματα. Θα πρέπει να φανούμε προσεκτικοί. Έτσι και αλλιώ νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι το 2013 είναι το έτος της ΚΕΠΑ. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στους συναδέλφους, λέει ο κ. θα θέσω τρεις ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά την παρέμβαση στο Μαλί, τη δύναμη για το Μαλί. Σε κάποια φάση είχε προβλεφθεί να υπάρξει μια διεύρυνση αυτού που συμβαίνει στον Νίγηρα, διαφορετικού τύπου αποστολή βέβαια, και εκεί έχουμε να κάνουμε με την κατάρτιση των δυνάμεων ασφαλείας, αλλά όχι του στρατού. Στο Μαλί το θέμα με τον στρατό είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό και δύσκολο. Και θα πρέπει επίσης να καλύψουμε και τις ανάγκες που εκφράζουν ήδη έντονα οι δυνάμεις ασφαλείας της χώρας. Λοιπόν, διαρωτώ με αν μια διεύρυνση της προσπάθειας που έχει ξεκινήσει ήδη στον Ήγηρα προβλέπεται. Τώρα, για τη Σομαλία. εφόσον οι συνθήκες ασφαλείας το επιτρέψουν, είπατε ότι θα εγκατασταθεί μια αποστολή στο Μογκαντήσου. Αυτό είναι κάτι το οποίο δέχονται όλα τα κράτη-μέλη ή μήπω υπάρχουν έντονες αμφιβολίες και δισταγμοί. Και τέλος, υποτίθεται ότι οι υπουργοί μίλησαν για το λεγόμενο pooling and sharing τον συνδυασμό δυνάμεων εν Εγώ παρατηρώ ότι σε ορισμένες από δηλώσεις υπουργών και αναφέρομαι στον Γερμανό Υπουργό ε, εκφράζεται ένας σκεπτικισμός και μια εχθρότητα απέναντι στην αρχή του pooling and sharing. Τι γίνεται, αυτές οι διαφωνίες, αυτές οι διαφοροποιήσεις έχουν εξεκαθαρίσει, έχουν κατασταλάξει στο Συμβούλιο ή μήπω πάντα θεωρούν όλοι ότι τελικά με το pooling and sharing με ένα μαγικό τρόπο θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε τους περιορισμούς και τις δυσκολίες. Κάτι το οποίο θα έδινε ουσία στην ίδια την προσπάθεια. Αυτά, ο κ. Γκάλερ έχει στήσει το λόγο πρώτος. Ευχαριστώ. Μιλήσατε για προτάσεις της Κομισιόν για την τυποποίηση και την εναρμόνιση. Η ε, αντίδραση των κρατών μελών ποια ήταν μετά την παρουσίαση της Κομισιόν, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άμα δεν συμφωνήσουν τα κράτη-μέλη δεν γίνεται τίποτε. Επίσης ε, είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι ικανή για δράση, να παραμείνει ικανή για δράση και ε, αναφέρατε και τους εθνικούς αμυντικούς σχεδιασμούς και είπατε ότι αυτούς πρέπει να τους μελετήσουμε. Καλό θα ήταν αυτό αν σημαίνει ότι προσεγγίζουμε την ιδέα μιας ευρωπαϊκής ε, αναθεώρησης ή επανεξέτασης της άμυνας. Πρέπει να δούμε τους αμυντικούς σχεδιασμούς. Και στην προετοιμασία για τη Σύνοδο Κορυφής είπατε ότι στην πρώτη φάση θα γίνουν και σεμινάρια και διασκέψεις. Δηλαδή να περιμένουμε ότι στην προπαρασκευαστική φάση θα συμμετέχει ε, καταλήλως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Merci, ε, Monsieur ο πρόεδρος μας σήμερα ε, δύο φορές έκανε αναφορά για το 2013 ότι είναι το έτος που θα δοθεί σημασία στην ΚΕΠΑ και πρέπει να δοθεί σημασία παρά τα πολιτικά ελλείμματα τα οποία όλοι διαπιστώνουμε ότι έχει. Ακούσαμε ιδιαίτερη προσοχή για το επιχειρησιακό κομμάτι που αναφέρεται στο Μαλί έγινε αναφορά για τους κινδύνους, για τις τρομοκρατικές ενέργειες που πιθανόν να προκύψουν, ότι ο στρατός χρειάζεται εξοπλισμό, τα κράτη-μέλη πρέπει να συμμετέχουν. Γίνεται μια συζήτηση στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών αν θα αναβληθεί, αν θα, αναλάβει η Κιανόκρανη, ότι πρέπει να υπάρξουν εκπαιδεύσεις σε όλα αυτά συμπυκνώνεται ένα συμπέρασμα ότι αναφέρονται σε χρόνο μέλλοντος. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Η επιχείρηση αυτή χρονοδιάγραμμα έχει για να υπάρξει έναν τέλος. Σκοτώνονται καθημερινά άνθρωποι. Τίθενται σε κίνδυνο άνθρωποι. Όποιοι και να είναι αυτοί. Θα υπάρξει μια συντονισμένη αντίδραση από τα κράτη-μέλη. Γιατί πολύ φοβούμε ότι το να διαπιστώνουμε αυτά τα προβλήματα δεν προσφέρουμε και την καλύτερη, αν θέλετε, ε, παρουσία ή ενισχύουμε την πολιτική αδυναμία που έχουμε. Οι Υπουργοί Άμυνας που συναντήθηκαν στο Δουβλίνο εξέφρασαν ένα σχεδιασμό, ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό και αποφασιστικότητα, γιατί εκτιμώ ότι και αυτό το ζήτημα θα παραμείνει, αν θέλετε, ένα ζήτημα που θα ταλαιπωρεί και βεβαίως την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη και βεβαίως εμάς σαν Επιτροπή Άμυνας. Χρειάζεται συντονισμός και με μία λέξη αποφασιστικότητα. Τι έχετε να πείτε. Merci, euh, Madame Thank you, Mr. President. Mr. thank you for... Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για την ενημέρωση. Να ρωτήσω κάτι που αναφέρατε. Ε, στην παρουσίασή σας, στην κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μαλί. Οι διεθνείς επεμβάσεις σκοπό έχουν πρωτίστως την προστασία του λαού του Μαλί. Ε, όμως δυστυχώς αναφέρεται ότι ε, εκτελέστηκαν ε, ε, από τις ένοπλες δυνάμεις, έγιναν βασανισμοί και σεξουαλική βία έλαβε χώρα ε, σε πλαίσια, στα πλαίσια αντεκδίκησης ε, από τις ένοπλες δυνάμεις που ενίκησαν και πολλοί πέθαναν σε μια επιχείρηση στο Μάλι. Εμείς θέλουμε να εφαρμοστεί το, να εφαρμόζεται το ανθρωπιστικό δίκαιο στο Μαλί, αλλά ως ομάδα πιστεύουμε ότι πρέπει να ε, παρακολουθήσουμε περισσότερα στο βόρειο, περισσότερο στο Βόρειο Μαλί τα ανθρωπιστικά δικαιώματα καθ' όλη την μεταβατική περίοδο και πρέπει να δώσουμε έμφαση στην εκπαίδευση και στα πλαίσια της αποστολής της ε, EUTM. Θα ήθελα τα σχόλιά σας εδώ. Um, Ευχαριστώ. Κύριε Ποπόφσκι, ε, να διευκρινίσω λίγο τι συζητήθηκε στην συνάντηση. Ε, νομίζω ότι συμφωνήθηκε να συζητούνται αμυντικά θέματα ε, με κάπως χαλαρό τρόπο. Και πρώτη φορά ετέθη το θέμα αυτό ως πρόταση. Τι ακριβώς συμφωνήθηκε και ποιοι θα συμμετέχουν στις συζητήσεις αυτές, αν αυτές γίνονται. Θα ήθελα να το διευκρινίσουμε το θέμα αυτό. Ο κύριος Ζέλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και σας πολύ κύριε Ποπόφσκι για την έκθεση. Μιλήσατε για την πειρατεία στην Σομαλία και στις αφρικανικές ακτές γενικότερα. Μια προκλητική ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Που ε, έλαβα από κάποιον υπεύθυνο στην επιχείρηση Αταλάντη που λέει ότι εδώ ε, καταπολεμούμε τα αποτελέσματα χωρίς να καταπολεμούμε τα αίτια. Ε, καταπολεμούμε την πειρατεία, αλλά δεν βλέπουμε το αίτιο. Που ποιο είναι το αίτιο? Ότι εν τω μεταξύ οι ακτές της Αφρικής Ε, έχουν πρόβλημα λόγω της ε, υπεραλίευσης από τους ε, στόλους των σκαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τώρα μπορεί η πειρατεία να μετατοπιστεί και σε άλλες περιοχές. Μπορεί λοιπόν να συνεχίσουμε την αποστολή επί χρόνια, αλλά δεν θα κάνουμε τίποτα αν δεν καταπολεμήσουμε τα αίτια. Εμείς έχουμε μεγάλη υπερρύθμιση, αν θέλετε, της αλληλείας στη... Ε, στα ευρωπαϊκά ύδατα. Αυτό όμως αλλάζει, η κατάσταση αλλάζει άρδιν όταν φύγουμε από την Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν και πρότυπα ασφαλείας για τους εμπορικούς στόλους, αλλά μαζί με τις αφρικανικές αρχές και τους ε, φορείς υπεύθυνους για την ανάπτυξη στην Ευρώπη θα πρέπει να μελετήσουμε πώς θα καταπολεμηθούν τα αίτια της πειρατείας αυτής. Υπάρχουν σχετικές σκέψεις. Euh, Κυρία κύριε Πρόεδρε, κύριε Ποβόφσκι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πολύ λεπτομεριακή αναφορά σας στη άτυπο Συμβούλιο Άμυνας που έγινε. Δεν πρόκειται για την πρώτη συνάντηση αυτού του είδους, αντιθέτως από ό,τι πιστεύουν κάποιοι συνάδελφοι. Τώρα, δεν ήθελα καταρχά να κάνω ερωτήσει, ήταν ενδιαφέροντα αυτά που ήταν και κατά πρώτο λόγο δεν νομίζω ότι ο ρόλο μας είναι να κάνουμε σχόλια, αλλά ακούγοντα εσά και του συναδέλφου σκέφτηκα το εξή. την ε, ευρωπαϊκή ε, λοιπόν ε, εξωτερική υπηρεσία μας που δημιουργήθηκε στα πλαίσια της εντολής της κυρίας έχουμε όλα τα θέματα άμυνας και αρμοδιότητας και ασφάλειας σε ένα άτομο. Αυτό δεν συμβαίνει σε κράτος. Στα κράτη-μέλη μας έχουμε υπουργό Εξωτερικών, Υπουργό Ευρωπαϊκών Θεμάτων και ξεχωριστά Υπουργείο Άμυνας. Διαρωτώ με λοιπόν. Κατά δική σας άποψη, αυτή η ασυμμετρία δημιουργεί πρόβλημα, ανοίγει νέες ευκαιρίες. Ποια είναι η άποψή σας. Θυμούμε ότι στο παρελθόν, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, με κάποιους ε, ενδιασμούς αντιμετωπίζαμε τα άτυπα συμβούλια άμυνα. Γιατί πολλέ φορέ δεν διαρωτώμεθα τι είδου αποφάσει θα μπορούσαν να έχουν πάλι και τι, σε ποια πράγματα θα μπορούσαν να έχουν συμφωνήσει. Δεν μα άρεσαν πάρα πολύ τώρα. Άλλαξαν τα πράγματα, προχωρήσαμε, πέρασε μια δεκαετία, έχουμε σήμερα πολύ πιο σοβαρές προκλήσεις. Άρα, ποια είναι η άποψή σας για αυτή την κατάσταση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντάρτμος τελικά. Ευχαριστώ. ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Πολλές ερωτήσεις και σχόλια θα μπορούσα να κάνω. Ε, μία όμως, ε, σε μία θα επιμείνω. Είπατε το εξής στην ομιλία σας. Είπατε ότι ο εθνικός αμυντικός σχεδιασμός των κρατών μελών πρέπει να εξεταστεί. Αυτό τι σημαίνει, μπορείτε να το διευκρινίσετε. Αυτό που νομίζω ότι σημαίνει είναι ότι είτε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή κάποιο συνδυασμό των δύο θα εξετάσουν τον αμυντικό σχεδιασμό των εθνικών κρατών. Και τι θα γίνει σε περίπτωση διαφωνίας με τις προθέσεις των κρατών μελών στον τομέα αυτών. Παράδειγμα, η Βρετανική κυβέρνηση τώρα δίνει μάχη για το αν το πρόγραμμα Trident για τα υποβρύχια θα το αντικαταστήσει. Αν το κάνει αυτό, θα μειωθεί η ικανότητα της ε, Βρετανικής κυβέρνησης να αναπτύσσει ταχαίως δυνάμεις όπως το Αφγανιστάν ε, και Ιράκ. Εγώ δεν είμαι ειδικό να πω αν είναι καλή ιδέα ή όχι. Ίσως ε, θα πρέπει ο κ. Βανόρδε να με βοηθήσει. Αλλά αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρήσει ότι όποια κυβέρνηση λάβει η Βρετανική κυβέρνηση για το πώς θα ε, κάνει τον μελλοντικό σχεδιασμό. Εάν εσείς ε, διαφωνήσετε, τότε τι θα γίνει, τι θα κάνετε, τι θα θελήσετε να κάνετε και τι αρμοδιότητες και εξουσίες έχετε για να κάνετε κάτι. Εδώ θα ήθελα μια διευκρίνηση. Η κυρία Γκόμες. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη κύριε Ποπόσκη που δεν ήμουν παρούσα. Δεν μπόρεσα να σας ακούσω, αλλά θα ήθελα παρόλα αυτά να υποβάλω δύο ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, Εάν οι Υπουργοί Άμυνας σε αυτό το ανεπίσημο συμβούλιο μίλησαν για τη χρηματοδότηση των αποστολών και ΑΠΑ, κυρίως για την αύξηση της ε, συμμετοχής σε αποστολές όπως αυτή για το Μαλή πράγμα που θα είχε διευκολυνθεί αν υπήρχε κοινωτική χρηματοδότηση, κυρίως για τις χώρες που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν σε ανθρώπινο δυναμικό, αλλά δεν έχουν τα κατάλληλα μέσα αυτή τη στιγμή. Και εάν συζητήσατε και για την αμυντική βιομηχανία, τι έχετε να μας πείτε για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε τους περιορισμένους πόρους που έχουμε σε όλα μας τα κράτη, δεδομένου ότι έχουν γίνει, όπως ξέρετε, μεγάλες περικοπές. Πώς μπορούμε όλα αυτά τα οποία λέμε στη θεωρία για το pull and share να τα κάνουμε πράξη. Ευχαριστώ. Κύριε Ποβόφσκι, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για όλες τις ερωτήσεις που μου κάνατε. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να απαντήσω. Αρχίζω με τις δικές σας ερωτήσεις για την UTM στο Μαλί. Την... Είναι μέρος του σχεδιασμού μας να το θεωρήσουμε ως ε, ε, παράταση της αποστολής η οποία υπήρχε σε θέματα κατά στην Ιγυρία. Αυτή τη δυνατότητα λοιπόν για την παράταση αυτής της μη στρατιωτικής ε, αποστολής με κατάρτιση αστυνομικών στρατιωτικών δυνάμεων στο Μαλί, από την Νιγερία στο Μαλί. Το προβλέπουμε. Έχουμε δύο αξιωματικού συνδέσμους, στο, έναν στο Μπαμάκο και προβλέπουμε άλλου δύο που θα μπορέσουν να αναλάβουν το θέμα αυτό. Δεν μπορώ να δώσω το χρονοδιάγραμμα, δεδομένου ότι όλα αυτά θα γίνουν Βεβαίω όχι κατά τη διάρκεια αλλά επιπροσθέτως πρέπει να πω ότι από το μέσο σταθερότητας έχουμε κινητοποιήσει μέσα για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τις διοκτικές αρχές του Μαλή χρηματοδοτώντας την αγορά ε, εξοπλισμού, ε, επικοινωνίας και οχημάτων. Αυτή είναι μια απόφαση που είναι προηγούμενη εβδομάδα η Κομισιόν. Τώρα, ε, αυτό το οποίο είναι στο Μαγκαντήσιο δεν είναι κάτι το οποίο θεωρείται σε διαφεσβήτηση. Έγιναν συζητήσεις στο παρελθόν και τα κράτη-μέλη απλώς ήθελαν να τους διασφαλίσει κάποιος ότι θα υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες προστασίας, ο κατάλληλος εξοπλισμός και η κατάλληλη κατάρτιση που πρέπει να ολοκληρωθούν στο Μαγκαντήσιο. Αυτό έχει γίνει, άρα προφανώς κάτι τέτοιο θα ολοκληρωθεί στο δεύτερο εξάμενο. Τώρα, το pulling and sharing, που έχει σχέση και με την τελευταία της κυρίας Γκόμες. Δεν πρόκειται για μαγικό ραδαβδάκι, όντως. Και δεν θα έλεγα ότι έχουν ενδιασμούς τα κρατημέλη, θέλουν να δουν αποτελέσματα. Άρα, σε πρώτη φάση θα καταλήξουμε στα συμπεράσματα όλου αυτού του εγχειρήματο φέτος, το δεύτερο εξάμεινο. Εάν θυμάσαι, τα κράτη-μέλη συμφώνησαν τον ε, κώδικα συμπεριφοράς που θα ακολουθήσουν για το pull and sharing για να μπορέσει να υπάρξει καλύτερη ε, διάρθρωση και διασύνδεση όλες αυτές τις φιλοσοφίες σε εθνικό επίπεδο. Χρειαζόμαστε όμως το κάποιο το πολύ πρόσφατο χρόνο ώστε να γίνει κάτι σε εθνικό επίπεδο πρώτα απ' όλα και μετά να δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα. Όπως προαναφέρθηκε, η συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο, στα επίπεδα αυτή τη φαίνεται ότι υπόσχεται πολλά και έχουμε πολλά επιτυχή αποτελέσματα τέτοιου είδους ε, ε συντονισμένης ε, ε, συνεργασίας σε επίπεδο Ολλανδίας-Βελγίου. Ε, Τώρα, ο κύριος Γκάλαχερ έθεσε κάτι για την τυποποίηση. Τέθηκε το θέμα για να μπορέσει να γίνει η ομαλή μεταφορά εξοπλισμού. Θα δώσω ένα γερμανικό παράδειγμα. Όταν συζητούσε η Γερμανία το θέμα της παροχής ελικοπτέρων για να υποστήριξει τους Γάλλους, ανακαλύφθηκε ότι έπρεπε να υπάρχει η κατάλληλη τυποποίηση. Δεν νομίζω ότι θα προτείνει κάτι η Επιτροπή δεν θα προτείνει καμία νομοθετική αλλαγή. Αυτό είναι σαφές. Το γνωρίζουμε. Αλλά πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Εάν θέλουμε να μεταφέρουμε εξοπλισμό και πρέπει να, είμαστε, να έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να είμαστε σε καλύτερο επίπεδο ε, διαδραστικότητα των δυνάμεων που διαθέτουμε σε αυτό τον τομέα στην Ευρώπη, θα πρέπει να το θέσουμε το θέμα. Τώρα, στην πρώτη ερώτηση του κ. Ντάρτμουρ. Εμείς δεν έχουμε αρμοδιότητες, δεν μπορούμε να πούμε στα κράτη-μέλη τι, τι να κάνουν. Απλώς θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι όταν τα κράτη-μέλη σχεδιάζουν να κάνουν κάτι, πρέπει να το κάνουν συντονισμένα. Δεν μιλούμε για θέματα τα οποία δεν είναι θέματα αρμοδιότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κάνουμε για κάποια θέματα σε θελούσια βάση για να βοηθήσουμε. Δεν παρεμβαίνουμε στον ε, αμυντικό σχεδιασμό του ΝΑΤΟ. Εάν θέλουμε όμως να προχωρήσουμε, ο κύριος Γκάλερ ανέφερε θέματα, αναθεώρησε θέματα στις άμυξες, μπορούμε να το κάνουμε. Δεν μπορούμε όμως και δεν θα οθήσουμε να κάνουν τίποτα τα κράτη-μέλη που δεν το θέλουν. Στα πλαίσια του pooling and share θα δούμε αν μπορούμε να θέσουμε από κοινού μεσότερε δυνατότητε που θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν ενδεχομένω και να είναι αποφελή και την Ευρωπαϊκή Ένωση και για το ΝΑΤΟ. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν στεγανά σαφή μεταξύ των δύο. Αν μπορέσουμε λοιπόν να αναπτύξουμε αυτέ τι κοινέ δυνατότητε, το κάνουμε με απόλυτη διαφάνεια και μεταξύ του ΝΑΤΟ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και του Γενικότερου Ευρωπαϊκού Επιτελείου. Το μήνυμα που μπορώ να μεταφέρω εγώ στα διάφορα κράτη-μέλη που οργανώνουν τέτοιου είναι ότι ό,τι γίνεται, γίνεται προς όφελος αμοιβαίο. Η ερώτηση του κ. Σοφοκλέους για την κατάσταση στο Μαλί. Σήμερα τα χρονοδιαγράμματα θα αρχίσουμε την ε, ε, αποστολή της εκπαίδευσης αυτή κάποια στιγμή Μάρτιο. Πρίλιο. Φαίνεται ότι θα παραμείνουμε εκεί για 15 μήνες, αλλά ίσως να χρειαστεί να παραταθεί η χρονική αυτή περίοδος. Και εκ παραλλήλου παρέχουμε και οικονομική υποστήριξη στην αφίσμα, στην Αφρικανική δύναμη η οποία έχει αναπτυχθεί στο Μαλί και στις γειτονικές χώρες, που θα είναι η βάση για τις νέες επιχειρήσεις, μελλοντικές επιχειρήσεις και ανοκράνων. Χρηματική λοιπόν υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διοικητική υποστήριξη και εξοπλισμός από τα κράτη-μέλη. Η κυρία Κοπά έθεσε το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό είναι μέρος της ε, εντολής της UATM, του Μαλή. Ανέφερα ότι θα υπάρχει έλεγχος, εποπτεία, επιτήρησης και μέλος της ε, εντολής της ε, αποστολής αυτής, αυτής της αποστολής στο Μαλή είναι και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα ανθρωπινιστικά. Δεν πρόκειται λοιπόν για την συνήθη στρατιωτική κατάρταση ε, κάποιων ε, στρατιωτικών ομάδων. Προβλέπουμε εκπαίδευση κατάρτιση και για θέματα ανθρωπιστικά και ανθρωπινών δικαιωμάτων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε και θέματα ε, Άμυνα στο παρελθόν, ακόμη στη δεκαετία του 80 και πήρε από την απόφαση πέρσι ο κύριος Βον Ρομπάι πριν από τη διάσκεψη κορυφής του ΝΑΤΟ στο Σικάγο το θέμα της άμυνας να το θέσει και στην μίληση διάταξη των συζητήσεων του ε, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αλλά βεβαίως οι αρχή κρατών και κυβερνήσεων θα το συζητήσουν το θέμα αυτό το Δεκέμβριο και η συνάντηση την οποία σχολίασα δεν ήταν η πρώτη, αλλά το πρώτο βήμα, αν θέλετε, για την προπαρασκευαστική αυτού του ε, Συμβουλίου. Κύριε Στέλλας, βεβαίως ε, ξέρουμε πολλές φορές ότι ε, σε θέματα πειρατείας πολλές φορές η οργάνωση προέρχεται από, την, από δυνάμεις, από την ξηρά. Έχουν μειωθεί όλες αυτές οι πειρατικές επιδρομές. Αλλά ξέρουμε ότι κυνηγώντα τους πειρατές στη θάλασσα δεν πρόκειται να σταματήσει αυτό το φαινόμενο και να εκκριζωθεί. Το θέμα είναι να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε και περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Εδώ η αλλιευτική δραστηριότητα είναι το σημαντικό. Γι' αυτό έχουμε ακριβώς ξεκινήσει ένα πρόγραμμα έτσι ώστε να καταστούν πιο ανθεκτικές οι δραστηριότητες αυτές, να βοηθήσουμε επίσης την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων στο κέρας της Αφρικής και επιπλέον αυτών ξεκινάμε να παρέχουμε ειδική, εξειδικευμένη μάλλον κατάρτιση στις χώρες της περιοχής και στις Σεϊχέλες, όχι μόνο στη Σομαλία, αλλά και στην Κένια, Τανζανία, μακροπρόθεσμα. Θέλουμε να τους βοηθήσουμε να δημιουργήσουν την ακτοφυλακή τους μόνοι τους και να μην εξαρτώνται από τις ναυτικές δυνάμεις ε, του ΝΑΤΟ ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει μια δράση που ονομάζεται Νέστορ με έδρα το Τζιμπουτί. Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο είναι στη φάση εκκίνησης. Το θέμα της πειρατείας είναι κάτι το ιδιαίτερα κερδοφόρο οικονομικά σαν δραστηριότητα και αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Θαυμάζω τον εκπρόσωπό μας, τον Άβαρχο. Example the other saying that the, ransoms... Coach. Και μου έλεγε ένα παράδειγμα ότι τα λίτρα που πλήρωσαν το 2011 ήταν 150 εκατομμύρια δολάρια. Ενώ τα χρήματα, τα εμβάσματα που έστειλαν οι Σομαλοί του εξωτερικού στην χώρα ήταν ένα δις, ξεπερνούσαν το ένα δις. Συνεπώς υπάρχουν δηλαδή πόρια, άλλοι υπάρχουν άλλες δυνατότητες για την κάλυψη των οικονομικών αναγκών. Για την κυρία Νέιτς, σχετικά με την ασύμετρία αν είναι θετική ή αρνητική. Κοιτάξτε, εμείς συνδυάζουμε λειτουργίες και των Υπουργείων Ανάπτυξης και των Υπουργείων Εξωτερικών και των Υπουργείων Άμυνας. Δεν είναι ένα πρόβλημα αυτό. Απλά αποδεχόμεθα ότι εξαρτώμεθα πλήρως από τα κράτη-μέλη και από την πολιτική τους βούληση. Εμείς εργαζόμεθα με τα μέσα τα οποία μας διαθέτουν οι ε, χώρες. Μερικές φορές ε, το ίδιο πρόσωπο εκπροσωπεί τις ε, χώρες του και ήδη ας πούμε την προηγούμενη εβδομάδα. Σας ανέφερα αυτή τη συνάντηση που έγινε στο Δουβλίνο. Ε, ήταν η Υπουργοί Άμυνας, ήταν η Υπουργοί Ανάπτυξης και συζήτησαν τα θέματα του Μαλή. Ε, και υπήρξε μια διασταύρωση των δραστηριοτήτων και των συζητήσεων. Οι υπουργοί είδαν τα πράγματα ο καθένας από τη δική του πλευρά. Αλλά εγώ είχα την δυνατότητα να ενημερώσω και τους υπουργούς για τα θέματα της ανάπτυξης σε σχέση με την ΚΕΠΑ και να παρουσιάσω τον καρπό της συζήτησης αυτής και στους υπουργούς άμυνας. Συνεπώς λοιπόν υπάρχει πρόοδος μέσω του συντονισμού των ε, θεμάτων που είναι υποσυζήτηση με τρόπο οργανωμένο. Ελπίζω, εν πάση περιπτώσει, έκανα ό,τι μπορούσα να απαντήσω τα θέματα του προγραμματισμού και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε τοπικό επίπεδο. Για την κυρία Γκόμες, τέλος, δεν υπήρξε ε, ειδική συζήτηση για τα θέματα της χρηματοδότησης. Εμείς ε, για το Μαλί χρησιμοποιούμε τον μηχανισμό Ατενά Εμείς προσπαθούμε να βελτιστοποιήσουμε, αν θέλετε, ε, τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Περί αυτού πρόκειται. Το, το pooling and sharing αυτό έχει σαν στόχο. Θέλουμε να περάσουμε στην επόμενη ταχύτητα όμως, να προχωρήσουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα και να καταστήσουμε το πέρασμα αυτό ένα πραγματικό ρεφλέξ και όχι απλά μια κατεξαίρεση διαδικασία. Καλώς. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω τους Βρετανούς συναδέλφους που είναι παρόντες εδώ σήμερα ότι υπάρχει ένας Ευρωπαίος Επίτροπος που τους ενημέρωσε ε, για τα θέματα της άμυνας. Ε, ο κύριος Μπαρνιέ δεν ήρθε όμως εδώ, σας καθησυχάζω, ο στρατάρχης ε, του Βρετανικού στρατού αλλά ως υπεύθυνο για τις κοινέ προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς ε, κάναμε μία συζήτηση πριν λίγες μέρες σε σχέση με τις ικανότητες που έχουν οι στρατοί των κρατών μελών. Ε, είναι σαφές ότι όλα τα Υπουργεία Άμυνας προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τους πόρους που έχουν στη διάθεσή τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ανάλογα με τα μέσα που έχουν τα κράτη-μέλη, ανάλογα είναι και τα μέσα που διαθέτουν στους στρατούς τους. Ε, η αλήθεια είναι ότι όσο μεγαλύτερες είναι οι στρατιωτικές δυνάμεις, και αναφέρομαι εδώ στη Μεγάλη Βρετανία και την Γαλλία, οι περικοπές, οι δημοσιονομικές για τους δύο αυτούς στρατούς είναι ιδιαίτερα υψηλές και φοβάμαι ότι το μαλλί στην παρούσα φάση είναι το δένδρο το οποίο ε, κρύβει το δάσος αν θέλετε. Ανησυχώ λοιπόν για όλα αυτά τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν τον Ιούνιο του 2013. Έχουμε μεν μέλλον, βρισκόμαστε στο μέσα Φεβρουαρίου, αλλά δεν βλέπω να υπάρχει καμιά ιδιαίτερη κινητοποίηση. Έτσι και αλλιώ, λίγοι είναι οι υπουργοί που παίρνουν μέρος στις ανεπίσημες συναντήσεις. Οι εργασίες της Task Force στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκονται σε επίπεδο εμβριακό. Φοβάμαι ότι θα καταλήξουμε στην προθεσμία του 2013 έχοντας μείνει πολύ πίσω και οι προτάσεις μας δεν θα είναι συγκεκριμένες, τα αποτελέσματα δεν θα είναι τα αναμενόμενα και απλά θα καταλήξουμε σε έναν επιπλέον κατάλογο καλών προθέσεων και ευχών. Και έτσι δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις απειλές, δεν θα μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες και τα κενά και τις προτεραιότητες μας. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να διατηρήσουμε μια στενή επικοινωνία εμείς θέλουμε να έρθουμε σε επαφή και να δημιουργήσουμε ακροάσεις με κάποιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί πρέπει να είμαστε σε θέση να υπενθυμίζουμε το ποιες είναι οι προτεραιότητες σε επίπεδο και πά. Εφόσον πράγματι τα κράτη-μέλη θέλουν να δώσουν στην πολιτική αυτή την θέση που της ανήκει, τη θέση που της ανήκει σύμφωνα με τις συνθήκες δεν μιλάμε για τη φαντασίωση και τον ιδεαλισμό κάποιων βουλευτών. Ζητάμε όμως την επικύρωση και τον σεβασμό των συνθήκων που έχουν ε, υπογραφεί από τα 27 κράτη-μέλη. Λοιπόν, τι προθεσμίες, τι, τι σημαντικές ημερομηνίες έχετε μπροστά σας, κύριε Ποπόσκη. Έχουμε τις ετήσιες συνεδριάσεις της υπηρεσίας μας το μήνα Μάρτιο και μετά προετοιμαζόμαστε τον Μάιο για τη συνάντηση του Συμβουλίου στο Λουξεμβούργο τον Ιούνιο. Ελπίζω οι Υπουργοί να είναι παρόντες αυτή τη φορά. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα επανέλθουμε αύριο με τους κυρίους Μπίλτ και Σικόρσκι. Έχουμε επίσης αύριο το πρωί νωρίς τον Νεοζηλανδό Υπουργό Άμυνας μετά τον κύριο Μπίλντ, μετά τον κύριο Σικόρσκι. Οι συντονιστές παρακαλώ μόνο να παραμείνουν στην αίθουσα, Μόνο οι συντονιστές.